στην εισηγήτρια την κυρία Χάνιμπο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με μικρόφωνο, παρακαλώ. Θα ήθελα να ένα χαιρετισμό σε όλους σήμερα που έχουμε πρόβλημα τις γυναίκες γιατί μιλούμε για τις ε, ετούσες άσυλο και τις γυναικές πρόσφυγες οπότε θα πρέπει έτσι να δει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς οι οποίοι αναζητούν την ασφάλεια μέσα στα σύνορά μας τη σήμερα ε, ημέρα. Έχουμε πάρα πολύ ανησυχητικέ ανισότητε σε σχέση με το τι γίνεται σε κάθε κράτο μέλο, δηλαδή με το πώ διεκπεριώνουν τι αιτήσει ασύλου, ιδίω όταν μπαίνει και ο παράγοντα ε, φύλλο. Ε, οπότε οι γυναίκε που αναζητούν κάποιο άσυλο δεν έχουν καμία εγγύηση ότι θα υπάρχει κάποιο είδου συνέπεια και λογική στο το άσυλο γιατί πολλέ φορέ έχουν αντιμετωπίσουν κάποιε πολιτικέ οι οποίε δεν ανταποκρίνονται σε κάποια παραδεκτά πρότυπα γιατί οι κρατικέ πολιτικέ που αφορούν τα δύο φύλλα δεν υλοποιούνται. Οπότε με αυτή την έκθεση θέλουμε να προτείνουμε κάποιες νέες κατευθυντήριες γραμμές για να μπορέσουμε να άρουμε αυτά τα κενά της νομοθεσίας γιατί δυστυχώς είναι καθημερινή πραγματικότητα η βία για τις γυναίκες και τα κορίτσια που φεύγουν να γλιτώσουν τη βία και έχω ακούσει ε, αποτρόπες αφηγήσεις για κακοποίησεις και βία και βλέπουμε ότι αυτό που να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες η σεξουαλική κακοποίηση, η εκμετάλλευση σε κάθε φάση της διαδρομής τους, ακόμα και σε έδαφος ευρωπαϊκό. Οι γυναίκες αλλά και οι ανήλικες που έτουν άσυλο ε, αναγκάζονται να παράσχουν σεξουαλική υπηρεσίες για λόγους επιβίωσης, στην πορνεία, ε, μέσα σε ένα φορτηγό, σε ένα σκάφος οπότε βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι οι γυναίκες χρειάζονται εναλλακτικέ, ασφαλέστερες αυτά τα λέμε στην έκθεσή μας οπότε θα πρέπει να πιέσουμε ε, ούτως ώστε το σύστημα ε, χορήγησης άσυλου θα πρέπει να προστατεύει τις γυναίκες και οι γυναίκες πρόσφυγες, αυτές που ζητούν άσυλο, ε, αντιμετωπίζονται με ίσο τρόπο χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά όπως και όλα τα υπόλοιπα θύματα της ε, βίας. Τις τελευταίες μέρες ε, μάθαμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που είναι μια πάρα πολύ πλήρης ε, συνθήκη που καταπολεμεί τη βία κατά γυναικών. Οπότε έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε με περισσότερη ισότητα μεταξύ φίλων ε, τις διατάξεις τις σχετικές με το άσυλο και την ισότητα ε, και έτσι να καλύψουμε τα όσα χρειάζονται γυναίκες και κορίτσια. Είπαμε επομένω ότι θα πρέπει να βοηθήσει και το κοινοβουλίο μας για να κυρωθεί αυτή η συνθήκη. Μόνο 12 κράτη-μέλη ε, την έχουν κυρώσει τα υπόλοιπα 13 τίποτα. Θα πρέπει όμως επίσης να δούμε και, και κάπως πιο μακρόπονα γιατί πολλές φορές μιλούμε ότι οι πρόσφυγες είναι κάτι σαν ένα βάρος, ένας μπελάς που φέρνει μόνο επιβάρυνση στη χώρα που τους φιλοξενεί. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχουν οι κατάλληλες ε, επενδύσεις, αυτό δεν ισχύει μακροπρόθεσμα. Και όλοι γνωρίζουμε ότι οι πρόσφυγες πολλά μπορούν να προσφέρουν ε, μακροπρόθεσμα στις κοινωνίες μας, αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε σοβαρά, να έχουμε πολιτική κοινωνικής ε, ένταξης, που να τους αγκαλιάζουν όλους. Οι γυναίκες έχουν ε, συγκεκριμένες ανάγκες, δηλαδή θα πρέπει να καλυφθεί το θέμα το γλωσσικό αλλά και η προστασία των παιδιών τους. Θα πρέπει να συνταχθούν και στην ε, αγορά εργασίας και έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα κενά στην ε, απασχόληση εδώ και 30 χρόνια είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε την σύμβαση τη σχετική με τους ε, πρόσφυγες με ισότητα, το 1994 το είπαμε αυτό και επίσης είπαμε να λάβουμε υπόψη τις κρατήρες γραμμές ε, της ε, είπα τη για τους πρόσφυγες είπαμε ότι οι γυναίκες και οι ανήλικοι είναι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται να γλιτώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 55% του υπολογίζει ο ΟΗΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε πολιτικές για να καλύψουμε τι ανάγκε του. Χρειάζεται μια προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τη διαφορά των φύλων σε κάθε φάση του ταξιδιού που κάνουν αυτέ οι πρόσφυγε Να τι προστατεύουμε όπω το χρειάζονται και σύμφωνα με όσα προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, λέει ο πρόεδρο, να δώσουμε τη σκητάλη στην Επίτροπο την κυρία Γιούροβα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και τους κοιόδες εισηγητές που έχουν συνεισφέρει σε μια πολύ σημαντική έκθεση. Ήταν πραγματικά εξαιρετική δουλειά που έκαναν. Η έκθεση αυτή τονίζει μια πολύ σημαντική πτυχή της κρίσης της ε, προσφυγικής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα γυναικών, κοριτσιών που εγκαταλείπουν ε, τις αιστείες τους λόγω πολέμου, ε, λόγω βίας και νομίζω πως ε, τα όσα είπε η είπατε αρμοστεί ότι το 20% των όσων φτάνουν από τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο είναι γυναίκες και το 33% είναι παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διεθνείς υποχρεώσεις για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται. Εγώ στηρίζω απόλυτα τη γενικότερη σύσταση έτσι ώστε να δοθεί μια ασφαλής και νόμιμη οδός για όσους διώκονται δεν θα πρέπει οποιαδήποτε ε, πολιτική κατά της ε, παράτυπης μετανάστευσης να οδηγήσει σε έλλειψη προστασίας αυτών που το αξίζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους νόμιμους δρόμους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα θα καταθέσει προτάσεις σχετικές. Εμείς πρέπει με ενεργό τρόπο να εξασφαλίσουμε πως οι άρτια αφιχθέντες που χρειάζονται προστασία έχουν τη δυνατότητα και συμμετοχής και πλήρους ένταξης στις κοινωνίες μας. Η επιτυχία της ένταξής τους αυτής εξαρτάται και από τις προθεσμίες. Δηλαδή, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονα εμπόδια γιατί είναι πολλαπλά τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν και το θέμα αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η προστασία υπηρεσιών που θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διάφορα βήματα για να έχουμε καλύτερη ένταξη και αυτό θα κατατεθεί το Μάρτιο του 2016. Βέβαια, η οδηγία για την ισότητα θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Πρέπει να σας πω πως η συστράτευση των ε, κρατών μελών είναι σημαντική, γιατί έχουν τα κατάλληλα εργαλεία. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχουμε και το Ταμείο για την ένταξη των προσφύγων και για το άσυλο και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με καλύτερο τρόπο για να αντιμετωπίζουν και τις ειδικέ συνθήκες ε, που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Δηλαδή θα πρέπει να μην πέφτουν θύματα ε, σκλαβιάς, εκμετάλλευσης, βίας, να δώσουμε τη μάχη κατά του τράφικινγκ. Και για το θέμα αυτό παρουσιάσαμε πέρσι σχέδιο δράση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν φέτος θα προτείνουμε να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει τα σχετικά στοιχεία κατά του τράφικιν στην ατζέντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019. Θα ήθελα να σε πιστήσω την προσοχή και στις νομικές υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να ε, φροντίσουν έτσι ώστε να μην ε, πέφτουν θύματα ε, εγκληματικών ομάδων αυτές οι γυναίκες και δίνουμε τη μάχη κατά του τράφικινγκ γιατί θεωρούμε πως είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το έχουμε συζητήσει και στις επαφές που έχουμε με τρίτες χώρες. Εσείς ζητήσατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην συνθήκη στη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης και να καταπολεμάσει τη βία κατά των γυναικών. Με χαρά σας ενημερώνω πως την περασμένη εβδομάδα 4 Μαρτίου του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για την προσχώρηση στη σύμβαση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί ένα σφαιρικό εργαλείο για να αντιμετωπίσει αυτό το διαδεδομένο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών. Συμπερασματικά λοιπόν θα κλείσω λέγοντας πως η Ευρώπη θα συνεχίσει να προσφέρει προστασία σε όσους χρήζουν ε, ε, προστασίας και για όσες γυναίκες και κορίτσια ζητούν ε, καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει τα μέτρα αυτά που θα λάβουμε να είναι αμοιβαίε προσπάθειες οι οποίες θα προσφέρουν καλύτερη προστασία και μεγαλύτερη ένταξη στις γυναίκες πρόσφυγες της χώρας μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εκθέση σας αυτή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ματέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συνάδελφο Χάνιμπολ για την έκθεσή της. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό ότι σήμερα, τη μέρα της γυναίκας, προσπαθούμε να δούμε πώς θα ε, άρουμε τις ε, ανισότητες. Το 38% των άσυλων στην Ευρώπη είναι γυναίκες και ακριβώς γι' αυτό το λόγο βλέπω ότι η κυρία Χάνιμπολ στην έκθεσή της πολύ σωστά έχει παραπέμψει ε, σε μια καινούργια πολιτική ε, για το άσυλο που να έχει κάποια ευαισθησία για τις γυναίκες, για τα κορίτσια που ζητούν άσυλο γιατί θέλουν να γλιτώσουν από τη βία και από τον πόλεμο και μας χτυπάνε την πόρτα. Επίσης είναι πάρα πολύ σωστό ότι χρειάζεται ανθρωπιστική προσέγγιση στις πιο ευάλωτες κατηγορίες όπως οι ηλικιωμένες γυναίκες ή οι έγκυες ή τα πολύ μικρά παιδιά. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με κάποια σημεία του κειμένου. Εκεί που αναφέρονται οι διαδικασίες του ασύλου, η επανένωση οικογενειών, αλλά επίσης και το πώ θα υπάρχει νομική αρρωγή στις γυναίκες γιατί όταν χρειάζεται νομική προστασία κοστίζει πάρα πολύ άρα ε, έτσι θα πρέπει να θυμιστούν με αυτά οι εθνικέ πολιτικές και άρα να δούμε πώς θα ρυθμιστούν σχετικέ αρμοδιότητες πώ όπως και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που ασχολούμεθα με τις δημοκρατικές ελευθερίες ε, να υπάρξει εδώ για όλες τις πολιτικές της ε, Ένωσης. Εμείς ως ΕΛΚ θέλουμε να υπάρχει μια εναλλακτική πολιτική, να υπάρχει μια ανθρωπιστική προσέγγιση στην μεταναστευτική κρίση, να λαμβάνεται υπόψη το τι χρειάζονται ε, οι ανήλικοι αλλά και οι γυναίκες που κινδυνεύουν από κακοποίηση σε αυτή, τους, σε τη φάση ζωής. Οπότε θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη και από την Europol και από την Frontex. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει παραπομπή στο κείμενο για το ότι χρειάζεται να υπάρχουν διαδικασίες υποδοχής που να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της γυναίκας ε, υγειονομικά ε, επίσης να υπάρχουν ε, χωριστοί χώροι για να αναπαύονται χωριστά από τους άνδρες δεν έχω άλλο χρόνο τώρα κυρία Γκαρθία Πέρες Ευχαριστώ Πρόεδρε είναι πολλαπλές οι κρίσεις που έπληξαν τα τελευταία χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική, η κρίση του ευρώ, η κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά χωρίς καμιά αμφιβολία η προσφυγική κρίση είναι εκείνη που αυτή τη στιγμή απειλεί να καταστρέψει το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αξίες μας, την αλληλεγγύη, την δικαιοσύνη και την ισότητα. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του εξή είναι εκατοντάδε χιλιάδε οι άνθρωποι αυτοί που διασχίζουν τη Μεσόγειο και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεφύγουν από το λοιμό, από το θάνατο και από το φόβο και ένα τμήμα όλων αυτών των ανθρώπων είναι ακόμα πιο ευάλωτες γιατί είναι γυναίκες και κορίτσια, πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, το 55% των προσφύγων που φτάνουν τους τελευταίους μήνες στις ακτές μας είναι γυναίκες και κορίτσια. Γυναίκες που έχουν χάσει τα πάντα και χάνουν την αξιοπρέπειά τους, που θα πρέπει να εκδίδονται για να πληρώνουν ε, ε, ε, αυτό το εισιτήριο του ονείρου της Ευρώπης. Οι γυναίκες που τις βιάζουν και είναι θύματα των διακινητών και των μαφιόζων. Και δεν μπορούμε εδώ να συνεχίζουμε απαθείς, να παρατηρούμε την κατάσταση. Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε, γιατί ε, πρόκειται για την ίδια την αξιοπρέπεια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε πολιτικές ένταξης, παιδείας, υγείας, δημοσίων υπηρεσιών, πρόσβαση σε όλα αυτά τα συστήματα για να εντάσσονται οι άνθρωποι στην κοινωνία μας. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η λύση του προβλήματος δεν είναι να τους ξαναγυρίσουμε πίσω στην άλλη όχθη της Μεσογείου. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η ευθύνη της Ευρώπης πρέπει να είναι να λύσει αυτό το πρόβλημα, να λύσει την κατάσταση, αλλά είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που σήμερα περιμένουν από την Ευρώπη να τους υλοποιήσει το όνειρο αυτό. Και εμείς τι τους επιστρέφουμε, μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με τους εμπνευστές Ευρώπης. Ευχαριστώ. Έχετε μπλε κάρτα από την κυρία Άτκινσον. Ε, θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Και τα ίδια ακούσαμε σήμερα το πρωί. Ε, ήμασταν ε, στο ίδιο πρωινό για την Παγκόσμια Μέρα της γυναίκας. Δεν άκουσα τίποτα για τι Ισλαμικέ ιδέε, τι μουσουλμανικές ιδέε, και δεν μιλώ για τους ακραίου. Αυτά είναι ασύμβατα με το φεμινισμό σα και το φεμινισμό μου που δεν νομίζω να ενδιαφέρουν. Δεν θα πρέπει εμεί να προστατεύουμε τα δικά μα παιδιά και τι δικέ μα γυναίκε με αυτά που βλέπουμε από μουσουλμανικές αξίε, πριν αρχίσουμε να θέλουμε να εντάσσουμε περισσότερους μουσουλμάνους που 40-50 χρόνια δεν έχουν ενταχθεί στι κοινωνίε μα τώρα θα ενταχθούν. Διαφωνώ απολύτως με αυτή την ε, παραδοχή. Το Ισλάμ δεν είναι καθόλου ασύμβατο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πολυμορφία, ποικιλία ε, και υπάρχουν πολίτες, άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη που είναι μουσουλμάνοι πολίτες. Αυτό που δεν είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τέτοιες ακραίες απόψεις. Είναι απόψεις που αυτό που κάνουν είναι να διχάζουν και να χωρίζουν τους ανθρώπους που δεν είναι μόνο από τον Ισλαμισμό και το Ισλάμ αλλά και από άλλες θρησκείες κατά της ισότητας των δικαιωμάτων των προσώπων ανδρών και γυναικών. Αυτό ε, πλήττει την καρδιά της Ευρώπης. Η μυσαλλοδοξία, η αδικία και όχι η μία ή άλλη θρησκεία αλλά οι αξίες που καταστρέφουν αυτή την αρχή που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε ορισμένοι να συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το Ισλάμ. Το πρόβλημα είναι η μυσαλλοδοξία, η έλλειψη αλληλεγγύης και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ε, το εγχείρημα αυτό αφορά όλους και όλες μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φονστόρχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ συζητάμε τώρα ευχολόγιο ε, της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φίλων για τις γυναίκες πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κρίση θα πρέπει να παραμένουμε ε, με ανθρωπιά, δεν χωρά καμία αμφιβολία και με ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά τι ζητάει το ψήφισμα τώρα, μόνο για γυναίκες πράγματα. Ε, ασφαλή ε, δίωδο στα κράτη-μέλη και πρόσβαση. Άρα να περάσουν όλοι. Γιατί το λέω όλα αυτά. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Τίμερμανς, είπε πρόσφατα ότι 60% των προσφύγων δεν είναι πρόσφυγες των μεταναστών, είναι μετανάστες. Και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε οικονομικούς μετανάστες και προσφύγες. Η Επιτροπή Γυναικών δεν το θέλει. Μα αυτό είναι περιφρόνηση αν φέρουμε τόσο κόσμο ή τους προσελκύσουμε και τους αφήσουμε μήνες ολόκληρους σε διάφορα γυμναστήρια και τέτοια ε, και μετά να τους επιστρέφουμε πίσω. Η έκθεση αυτή είναι ένα ευκολόγιο που υπερβαίνει κατά πολύ ε, τη δικαιοδοσία της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των φύλων που θέλει να χειραγωγήσει και να αποδιαιτήσει τα κρατη και χάνει τελείω την πραγματικότητα. Και όπω με πολλές εκθέσεις τη Επιτροπή Γυναικών δεν μπορούμε παρά να απορρίψουμε και την παρούσα. Ευχαριστώ κύριε Φωνστόρ. Έχετε μπλε κάρτα του κυρίου Φρουντσούλητσα. Τη δέχεστε? Παρακαλώ. 30 δεύτερα. Ε, first of all, ladies and gentlemen. Πρώτα απ' όλα κυρίες και κύριοι θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ σε όλες τις συναδέλφους μια υπέροχη άνοιξη, μια όμορφη ζωή, υγεία, ευτυχία για την 8η Μαρτίου. Ας το ευχηθούμε σε όλες τις γυναίκες, σε όλα τα κορίτσια στον κόσμο. Και παράλληλα, επιτρέψτε μου να σας κάνω την εξής ερώτηση. Όλες αυτές οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερη προστασία. Έτσι δεν είναι, όπου και αν βρίσκονται ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους, την εθνική τους καταγωγή. Πρέπει να κάνετε ερώτηση, συνάδελφε. Δεν ήταν μπλε κάρτα αυτή, συνάδελφε. Αυτές τις ευχές για τις γυναίκες σήμερα θα μπορούσατε να τις είχατε δώσει σε κάποια άλλη στιγμή. Η μπλε κάρτα είναι για να απευθύνουμε ερώτηση σε προηγούμενο μιλητή. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δώσω για 30, δευτερο... για 30 δευτερόλεπτα στην συνάδελφο για να απαντήσει. Καταπληκτική ερώτηση και συζήτηση έγινε σήμερα Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας και βλέπουμε το τεράστιο ενδιαφέρον πόσες γυναίκες είναι παρούσες. Είναι τρει και ο κούκο. φαντάζεστε τεράστιο ενδιαφέρον, έχει συγκεντρώσει πλήθη εδώ μέσα. κυρία Μαγκέρικα Μλίναρ από του Φιλελευθέρου για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτέλους έχουμε μια έκθεση που είναι ισορροπημένη, που είναι γεμάτη και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε επειδή ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συνεργασία με την εισηγήτρια και με τους σκιώδες οι οποίοι αναγνώρισαν πως πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτες γυναίκες. Η ανθρώπινη μετανάστευση δεν είναι κάτι καινούριο αλλά αυξάνεται επειδή είναι όλο και πιο ευάλωτες οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες στο τράφικινγκ, στην εκμετάλλευση, στη βία. Κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν πως ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε την 8η Μαρτίου είναι από τις γυναίκες που ζητάνε άσυλο και από τις ε, γυναίκες ε, μετανάστριες να αφαιρέσουμε τα δικαιώματα στην υγεία, στην αναπαρογή υγεία, στην προστασία και ε, να περάσουμε σε μια πιο ταχεία διαδικασία οικογενειακής επανένωσης. Νομίζω ότι αυτό που μας περιμένει δεν είναι μια προσφυγική κρίση μια μεταναστευτική κρίση, αλλά μια προσφυγική κρίση και μια κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ συχνά τα δικαιώματα αυτά αγνοούνται από όλους και θεωρούνται μια λεπτομέρεια ή μια πολυτέλεια ή και μια άχρηστη επιπλοκή. Είναι δύσκολο να δούμε πολλές φορές την προοπτική του φίλου στα θέματα αυτά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ανεχθούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προστατεύει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Οι γυναίκες που αιτούνται άσυλο ζητούν συγκεκριμένη προστασία και ξέρουμε ότι σε πολλά κέντρα υποδοχής έχουμε ε, κακό φωτισμό δεν υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια για τις γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες ή για αυτές με οικογένειες ε, και επίσης είναι υπερβολικά γεμάτα. Άρα λοιπόν για να ακολουθήσουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε και τους λόγους της βίας κατά των γυναικών και εδώ θα συμπεριλάβω και το τράφικινγκ και τη σωματεμπορία για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό θα πρέπει στις διαδικασίες ειρήνευσης να εμπλακούν περισσότερο οι γυναίκες έτσι ώστε να επιληθούν οι σειράξεις οι οποίες αποτελούν και την ρίζα οποιασδήποτε οικονομικής κρίσης. Σας ευχαριστώ πολύ. η κυρία Μάριν ε, από την ΚΟΕ για ένα λεπτό παρακαλώ. Η 8η Μαρτίου μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε περισσότερο τους αγώνες των γυναικών, τους καθημερινούς. Και έτσι μπορούμε τώρα να αναδείξουμε και τα προβλήματα των ε, προσφύγων και των εντουσών άσυλο. Επίση θα πρέπει να υπάρχει ασφαλής διέλευση, θα πρέπει να υπάρχει πανένωση οικογενειών, αλλά ακριβώ επειδή είναι πιο ευάλωτε οι γυναίκες, ακόμη περισσότερο χρειάζεται αυτή η προστασία. Χρειάζονται επομένω κάποιε τέτοιε ανθρωπιστικέ διαδρομέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε στα σύνορα που είναι οι γυναίκε και οι συνθήκε εκεί είναι απαράδεκτε τώρα όσον αφορά την επανένωση των οικογενειών, μια σειρά χωρών ε, με παράδειγμα τρόπο αντιμετωπίζουν αυτή την αρχή, αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι χτύπημα στην οικογένεια αλλά κυρίω στους ανηλίκους και στις ε, γυναίκε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επομένω να μπορούν να επανενωθούν οι οικογένειε και συμφωνώ με όλα όσα λέει η έκθεση αυτή. Είναι κρίμα που δεν ισχύει το ίδιο με δεξιά και με του ε, ρατσιστέ. Έχετε κάποια επερώτηση από την κυρία Γουίνμπεργκ. Αποδέχεστε. Ναι, λέει η κυρία Μπιόρκ. Μισό λεπτό. Δυστυχώς έχουμε τόσους νέους μετανάστες που επί σε σεξουαλικά, που βιάζουν. Είδατε τι έγινε το 2015 στην Κολονία και στην Στοκχόλμη. Είδαμε ότι τα κουκούλωσαν οι αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για μια μάστιγα. Θα πρέπει επομένως να υπάρξουν εγγύησεις ασφάλειας. Και για τι γυναίκε τη Δύση όμω, θα πρέπει να είναι δυνατόν και οι γυναίκε τη Δύσης να μην πέφτουν θύματα τέτοιες ενέργειες. Η κυρία Μπιόρκ. Ναι, ναι, κλασική αντιμετώπιση αυτή. Ε, φαίνεται απέναντι και αντιπάλους τον έναν άνθρωπο απέναντι στον άλλο δεν είναι έτσι. Αυτό που λέτε είναι υποκριτικά. Το μόνο το οποίο κάνετε είναι να διατυπώνετε τους ισχυρισμού και ρατσιστικού πρόεδρου. Ε, ο κύριο Φουρτάσον για 1,5 λεπτό από του Πρασίνου. Ευχαριστώ. Χθε. Ήταν άλλη μια επέσχυντη μέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ειδωμένη χιλιάδες γυναίκες και παιδιά ε, ε, ε, διανυκτέρευαν στη βροχή και στη λάσπη σε ελεηνές συνθήκες. Τι γινόταν στη Σύνοδο Κορυφής. Να παραβιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, να προωθηθούν οι ε, συλλογικές απελάσεις και επιστροφές αντί να γίνεται, όπω λέει ο ατομική εξέταση της κάθε περίπτωση. Βλέπουμε τι κάνουν οι κυβερνήσεις. Άλλη μια ε, μαύρη πενταετία της ένταξης. Θα εγκρίνουμε τώρα την έκθεση Hannibal, την οποία θέλω να ευχαριστήσω για την εργασία τους, με πολιτικές που ζητούμε και συστήνουμε για να προστατεύονται γυναίκες πρόσφυγες. Καλό θα ήταν για αλλαγή οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσουν τι τους λέμε. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει η βία, σεξουαλική, η εκμετάλλευση, οι εκβιασμοί ε, είναι να αλλάξει πολιτική για τους πρόσφυγες. Χρειαζόμαστε ασφαλείς οδούς. Μόνο έτσι θα καταπολεμήσουμε τη διακίνηση ανθρώπων και γυναικών. Ε, να προωθήσουμε την οικογενειακή επανένωση. Οι γυναίκες να έχουν δικαίωμα να κάνουν ξεχωριστή αίτηση ασύλου εκτός ε, του συζύγου. Διαφορετική ε, προστασία στις θυλάζουσες μητέρες, τα παιδιά βοήθεια ψυχολογική στι γυναίκες που υπέστησαν ε, βία, σεξουαλική κλπ. Όλα αυτά είναι τα πιο θεμελιώδη, τα πιο βασικά δικαιώματα των γυναικών. Ακούστε μα επιτέλου κάποια φορά για αλλαγή, κάποια από αυτά που σα ζητάμε κάντε τα. Ευχαριστώ. Κύριε Ουρτάσον, έχει μπλε κάρτα. Κυρία Άτκινσον, τη δέχεστε. Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, από την ομάδα της η κυρία Γιούτο για ένα μισή λεπτό. <clears throat> Αγαπητοί συνάδελφε, ως πολίτες αλλά και ως θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, καλούμεθα να αποκτήσουμε αυτή την τεράστια πρόκληση. Έχουμε όλου αυτού του ε, πρόσφυγε αυτού του εντός άσυλο, χτυπάνε την πόρτα και έχουμε πάρα πολλέ γυναίκε και πάρα πολλά παιδιά που είναι για πρώτη φορά η πλειοψηφία και αυτό δεν είναι όμω κάτι που συνέβη τώρα για πρώτη φορά αλλά έτσι έχουμε τώρα μια αλλαγή δημογραφική. Έχουν πάρα πολλές αιτίε. Έχουμε τόσες ένοπλε συγκρούσεις στις χώρες προέλευσης. Έχουμε ε, τόση, τόση βία έχουμε καταπάτηση των δικαιωμάτων αλλά έχουμε όμως ανετία και τις κλιματικές ε, αλλαγές έχουμε την καταχρηστική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δεν θα, θα πρέπει να μείνουμε αδρανίστια της, είμαστε συνυπεύθυνοι θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και να κάνουμε κάτι για αυτή την κρίση ε, βλέπουμε πόσο υποφέρουν οι γυναίκες από αυτή την κρίση και άρα τι θα κάνουμε πρώτα πρώτα να μείνουμε άνθρωποι χρειάζεται με συγκεκριμένο τρόπο έκφραση έκφραση αλληλεγγύης. Χρειάζεται υποδοχή, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και από τα 28 κράτη-μέλη και έτσι μπορούμε, θα μπορούμε να ανασχέσουμε ε, αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Δεν θα πρέπει ο, ο καθένας να κλείνεται, να κλείνει τα σύνορά του ε, και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και σε κάποιες χώρες σαν την Τουρκία που έχουν κάποια διαφορετικά πρόβλημα από αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει χρόνος που μπορούμε πια να χάσουμε και άρα θα πρέπει να υπάρχει νομική υποστήριξη ε, και οπότε θα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι γυναίκες φεύγουν από το σπίτι τους και τρέχουν διατρέχουν τους κινδύνους και αυτές και τα παιδιά τους. Η πρόεδρος. Έχετε μπλε κάρτα από την ίδια ομάδα, δεν, δεν ε, δέχομαι κάρτα από την ίδια σας την ομάδα να γίνει ερώτηση. Α, Α, μου είπαν ότι είστε από την ίδια ομάδα. Από άλλη ομάδα είστε. Τη δέχεστε. Της κυρίας Άτκινσον. Παρακαλώ. 30 δεύτερα. Ε, ένας από του λόγου που δεν είμαστε στην ίδια ομάδα είστε εσεί. Ακριβώ. Γιατί έχετε μια προσέγγιση προ το σοσιαλισμό και του Πρασίνου που με οδήγησαν να φύγω από την ομάδα σα. Δεν κάνετε καμία διακρισία ανάμεσα στου οικονομικού μετανάστε και εκείνου που είναι γνήσιοι πρόσφυγε. Και πάλι στην ομάδα σα υπάρχει διάσταση απόψε ότι κάνετε αυτή τη διαφορά ή όχι. Ποιο είναι οικονομικός μετανάστης και ποιος πρόσφυγας. <coughs> Ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Όχι, δεν υπάρχει καμία διαφορά το να προσπαθεί κανεί να γλιτώσει τον ε, θάνατο. Γιατί ε, όταν κανεί φεύγει, τρέχει μακριά από έναν πόλεμο, θέλει να επιβιώσει και δεν μπορεί ούτε να γλυρίσει τη γη ή επειδή έχει κάποια δικτατορία που τον κυβερνάει όλα, αυτές, όλα αυτά που λέτε είναι διχαστικά σαν διακρίσεις είναι πράγματα που καθόλου δεν τα έχει ανάγκη η Ευρώπη Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Ντορνανό ε, από την ομάδα της για ένα λεπτό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Μόλις επέστρεψα από το Ιράκ όπου σε μια ανθρωπιστική αποστολή επισκέφθηκα τους χριστιανούς που τους διώκουν και τους καταδιώκουν οι Ισλαμιστές. Δεκαετίες αγωνίζομαι υπέρ των γυναικών και της ε, εξωπρέπειάς τους στην Ευρώπη και τώρα ε, έκθαμβη ε, και όλα απορία βλέπω την έκθεση της συναδέλφου. Ε, δεν υπάρχει καλύτερη έκφραση του ελευθεριάζοντος σοσιαλισμού τελείως αποσυνδεδεμένο από την πραγματικότητα. Πού είδατε ότι οι γυναίκες ζητάνε άσυλο επειδή είναι ε, ε, θύματα ΛΟΑΔ. Ε, πού είναι αυτά, ε, τι ε, αστικά κριτήρια της Δυτικής Ευρώπης με φλου έννοιες και άσχετες αυξάνεται τον κίνδυνο μιας πιο μαζικής ακόμα μετανάστευσης. Πώς αποδεικνύεται ότι κάποιος είναι θύμα ε, λόγω ε, ε, της υποτιθέμενης διεμφυλικής τους ιδιότητα και πώς τεκμέρεται αυτό, τι πιστήρια θα απαιτήσετε ως Ευρωπαία γυναίκα πραγματικά με θλίβει ο τρόπος με τον οποίο διαστρέφεται τα πράγματα και τα χρησιμοποιείτε ονόματι της ηθικής σας δικτατορίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιέζει ο χρόνος λέει Πρόεδρος και τώρα έχω επιτρέψει μπλε κάρτε προ του εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων το εξή δεν θα το δεχτώ, στο λέω από τώρα για να μην απογοητευτείτε που δεν θα σα δίνω το λόγο. Η επόμενη ομιλήτρια τώρα είναι η κυρία Κωνσταντ Λουιγκρίπ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να αφιερώσει αυτή την ημέρα στο θέμα των γυναικών. Των γυναικών προσφύγων, των γυναικών που αιτούνται άσυλο, των πολύ αριθμό παιδιών που τη συνοδεύουν. Και εδώ στην αίθουσα καμία πολιτική ομάδα και κανείς ε, βουλευτής και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μην δείξει ευαισθησία για αυτόν τον ανθρώπινο πόνο, για την οδύνη που φαίνονται και φτάνουν συνέχεια στα ευρωπαϊκά σύνορα. Μιλώ για την κατάσταση των γυναικών προσφύγων ε, που ετούνται άσυλο στα διάφορα σημεία της Ευρώπης. Εμείς στο ΕΛΚ επειδή έχουμε μπροστά μας την έκθεση Hannibal, θέλουμε να προτείνουμε ένα εναλλακτικό ψήφισμα, γιατί δεν θέλουμε να συμφωνήσουμε 100% με όσοι συμπεριλαμβάνει η έκθεση Hannibal. Έχουμε λοιπόν ένα εναλλακτικό ψήφισμα, το οποίο θα εστιάζει στις προτάσεις, οι οποίες θα είναι αξιοπρεπείς, ανθρώπινες, αλλά και ρεαλιστικές και υπεύθυνε για το θέμα της υποδοχής των γυναικών προσφύγων και των των ασυλών. Θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές, λογικές, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες με συγκεκριμένες διαδικασίες για να ξεπεραστούν, για παράδειγμα οι ανάγκες γυναικών επαναλαμβάνω με ρεαλιστικό τρόπο και θα θέλαμε ως πρώτη προτεραιότητα να θέσουμε τη μάχη εναντίον οποιοδήποτε τράφικη ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης που γίνεται από τα δίκτυα της μαφίας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρία Γενά, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ένα τρίτο Τόν ε, τον ετούν τον άσυλο σήμερα είναι γυναίκες. 38% των μεταναστών στην Ευρώπη είναι γυναικόπαιδα. 55% των αφήξεων στην Ελλάδα σήμερα είναι γυναικόπαιδα. Τι μας δείχνουν αυτά τα στοιχεία, Τι συνθήκες που επικρατούν που είναι απάνθρωπες και στις χώρες προέλευσης και καταγωγής και με πολέμους και όλες τις καταστάσεις αστάθειας που επικρατούν. Αλλά μας δείχνουν και ιδιαίτερα ότι για τις γυναίκες η βία με βάση το φύλλο είναι μεγάλη. Η Ναγουάν Σουηφή ήρθε την περασμένη εβδομάδα ε, να μας καταθέσει τη μαρτυρία της για τις δραματικές καταστάσεις που ζουν αυτές οι γυναίκες. Μας δείχνουν τα στοιχεία αυτά επίσης πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες της κατάστασης της γυναίκας αυτής. Πρώτον, με βάση το φύλλο, όταν ζητούν το καθεστώς του πρόσφυγα, το καθεστώς αυτό ε, και η σύμβαση έχει συνταχθεί από άντρες για άνδρες και χρειάζεται επιγόντως αναθεώρηση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες των γυναικών ε, κατά τη μετανάστευση. Ας πούμε, ο γενετικός ακροτηριασμός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πολύ πιο σοβαρά. Επίσης, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες υποδοχής για να έχουν πρόσβαση και στην αναπαραγωγική υγεία οι γυναίκες και στην άμβλωση με ασφάλεια. Επίση, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να ενταχθούν οι γυναίκε αυτέ στην κοινωνία για να μπορούν να ζουν στην Ευρώπη. Αν δεν κάνουμε τίποτα να δρανίσουμε, η ιστορία θα καταγράψει ότι η Ευρώπη μαζικά ε, αφίσταται από τι αρχέ τη ουμανισμό, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλεγγύη. Αυτό ζητεί η παρούσα έκθεση και επ' ευκαιρία θέλω να συγχαρώ την Μέρη Χάνιμπολ για την εξαιρετική τη εργασία. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Βυσνιέσκα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα οποία ακούγονται για την κατάσταση των γυναικών προσφύγων είναι καταθλιπτικά. Και καμιά φορά διαπιστώνουμε ότι τελικά χρειάζεται να εκπορνευθούν για να καταφέρουν να φτάσουν στην Ευρώπη και όχι μόνο πριν ξεκινήσουν αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους και σε όλο αυτό το ταξίδι αντιμετωπίζουν βία, είναι πολύ άσχημες οι συνθήκες στα κέντρα υποδοχής και αυτό οδηγεί σε όλο και περισσότερες τραγωδίες. Τώρα, άσχετα με το τι πιστεύει ο καθένας μας για την κρίση αυτή, βλέπουμε πως η κατάσταση απαιτεί μία άμεση απόκριση για να βελτιωθεί η τύχη και η ζωή αυτών των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δυστυχώς, για μια φορά ακόμα και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύεται πως δεν μπορεί να σταθεί ενωμένο και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουν κάποια άλλα θέματα. Ε, δεν νομίζω ότι θα πρέπει εδώ τα δικαιώματα τύπου ε, αμβολώσεων θα πρέπει εδώ να μας ε, ε απασχολούν. Επόμενη μιλήτρια η κυρία Μπεσέδα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδιάς την κυρία Χάνεπουλ για μια εξαιρετική έκθεση. Είναι πλήρης και έφτασε και την κατάλληλη στιγμή. Είναι πολύ επίκυρη γιατί έχουμε το φαινόμενο αυτό το πολυδιάστατο το οποίο όλο και εξαπλώνεται. Έχουμε την παράλυση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που δεν μπορούν να δώσουν τη μοναδική απόκριση που αξίζει, που είναι μια κοινή πολιτική ασύλου και έχουμε και κάτι που έχει αλλάξει στην κρίση των προσφύγων. Έχουμε καταρχήν την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει καταρρεύσει και που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ανθρωπιστική κρίση μέσα στο ίδιο της στην επικράτεια και έχουμε και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει 700 εκατομμύρια σε βοήθεια. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι παραπάνω από τα μισά άτομα που φτάνουν είναι γυναίκες και παιδιά, όχι άντρες πρόσφυγες. Άρα λοιπόν μιλάμε για τεράστιο εκτοπισμό πληθυσμών που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι γυναίκες και οι άντρες ε, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά οι γυναίκες, τα κορίτσια ε, αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα, ε, βία. Χτες μας είπε ο κύριος Τούσκ πως μπορεί το θέμα, ότι το θέμα έκλεισε. Ναι, βέβαια. Αλλά η λαθρομετανάστευση δεν σημαίνει πως κάποιοι που έχουν ε, δικαίωμα σε άσυλο δεν θα πρέπει να απολαύσουν το δικαίωμα αυτό όπως λέει η Σύμβαση της Γενέβης, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης την οποία σύντομα θα υπογράψουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κούνεβα παρακαλώ για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. χρόνια πολλά σε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες που συνεχίζουν να παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Φαίνεται ότι το Στρασβούργο από τις Βρυξέλλες δεν, μόνο, δεν τα χωρίζουν μόνο 440 κιλόμετρα αλλά μια άβυσος. Ενώ εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε μια έκθεση που ζητάει να προστατευτούν με ανθρωπιά οι γυναίκες πρόσφυγες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες λέει ότι καλώς έκλεισαν τα σύνορα η Αυστρία και οι άλλες χώρες και κάποιες κυβερνήσεις περνάνε ανοιχτά στο ρατσισμό λέγοντας ότι δεν δέχονται μισογουμάνους στο έδαφο, τους. Ενώ εμεί ζητάμε ασφαλείς και νόμιμους δρόμου για πρόσφυγε και μετανάστες το Συμβούλιο κάνει ένα απάνθρωπο παζάρι με την Τουρκία για κάθε γυναίκα πρόσφυγα που τα περνάει τα παίρνει άσυλο μια μετανάστρια τα αποχρεώνεται να επιστρέψει στην Τουρκία. Έχει δίκιο η υποτιαρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες όταν λέει ότι μια τέτοια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία μπορεί να είναι παράνομη γιατί τα παραβιάζει και το διεθνώ και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σα καλώ να ψηφίζω με την έκθεση τη συνάδελφου Χάιν. Με την έκθεση, με τη σκέψη να στηρίξουμε τα δικαιώματα των προσφύγων. Τελείωσε ο χρόνος σας. Ένα λεπτό είχατε μόνο, κύριε Κούνεβα. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερο χρόνο. Είχατε ένα λεπτό μόνο. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Ράιντκε, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι. Πάνω από 150 χρόνια πριν είχαμε κάποια αγοριστή που είχε πει πόσο προβλήματα υπάρχουν όσον αυτά τα δικαιώματα των γυναικών, των ε, έγχρωμων, των ε, λεσβιών και σήμερα αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συζητούμε την πατριαρχική βία, την καταπολέμηση της βίας και των γυναικών. Γιατί υπάρχουν κάποιες πτέρυγες στο κοινοβούλιο που δεν θέλουν να γνωρίσουν ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδων γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μέσα στην Ένωση πρόσφυγες ίδιες και βλέπουμε ότι και αυτές χρειάζονται προστασία. Γιατί θα πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμό μεταξύ κάποιων να χρειάζονται και κάποιε να μην χρειάζονται. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει το Κοινοβούλιο. Είναι παγκόσμια τα γυναικεία δικαιώματα. Δεν περιορίζονται από κατηγοριοποίηση εθνοτική ή από σύνορα ή από θρησκεία. Θα πρέπει να προστατευτούν οι γυναίκες. Αλλά επίσης θα πρέπει ο φεμινισμός να στηριχτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η απο συνορα η απο θρησκεια θα πρεπει να προστατευτουν οι γυναικε αλλα επιση θα Πάρκερ, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ε, ένα point system όπως η Αυστραλία για να ελέγχει τη μετανάστευση θα μπορούσαμε να προστατεύουμε καλύτερα τους πρόσφυγες. Αλλά επειδή έχουμε 300.000 που έρχονται το χρόνο στη Βρετανία ε, προσπαθεί ε, η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις ανησυχίες του κόσμου που θεμητές είναι δεν μπορούν να έρχονται ανεξέλεγκτα, ανειδίκευτοι ε, ε, άνθρωποι χωρίς να ελέγχουμε και το ποινικό τους μητρό. Πάνω από ένα εκατομμύριο ήρθαν στην Ευρώπη το 2015. Λέει η κυρία Μέρκελ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθαρρύνει ευάλωτες γυναίκες και παιδιά να ε, κινδυνεύουν στη Μεσόγειο για να πέφτουν στα νύχια των διακινητών και να χάνουν τη ζωή τους. Η Ευρωπόλ λέει ότι 10.000 παιδιά ε, αγνοούνται και πολλά έχουν μπλέξει και σε κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει τις θύρες σε εκατομμύρια πολίτες από χώρες που θεωρούν τις γυναίκες πολίτες δεύτερης κατηγορίας για να μην πούμε για τους ΛΟΑΔ. Ε, είδαμε τι έγινε στην Κολονία και τη Σουηδία την πρωτοχρονιά με επιθέσεις σεξουαλικού περιεχομένου και εξευτελιστικού για τις γυναίκες. Για να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες θα πρέπει να καταργήσουμε αυτές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπονάνο, για ένα λεπτό Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας διαβάσω κάτι. Για να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Κάτι το τόσο σημαντικό. Προσέξτε να μην κάνετε μια γυναίκα να κλάψει γιατί στα δάκρυά της κρύβεται ο Θεός. Βγήκε από την πλευρά του άντρα η γυναίκα. Ούτε βγήκε από τα πόδια, ούτε βγήκε από την κεφαλή, ούτε κατώτερη ούτε ανώτερη. Βγήκε από το πλευρό του. Γιατί είναι και για να είναι ίση. Ε, για να προστατεύεται. Εκεί κοντά στο ε, μπράτσο του, κοντά στην καρδιά, για να την αγαπάει. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το σκεπτόμαστε. Αυτό θα πρέπει να εφαρμόζουμε για τις γυναίκες λιγότερη υποκρισία και περισσότερες πράξεις να λέμε λιγότερα λόγια και περισσότερες σοβαρές πράξεις. Η κυρία Γκάλ Πέλτς για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε σε αυτήν την Παγκόσμια Μέρα για την Γυναίκα συζητούμε για την βία κατά των γυναικών και για τις ε, γυναίκες μετανάστερες. Σίγουρα και οι γυναίκες και τα παιδιά προσπαθούν να γλιτώσουν από τον ε, πόλεμο ελπίζουν σε μια νέα καλύτερη ζωή στην Ευρώπη και σε αυτό το ταξίδι είναι εκτεθειμένοι στην ε, βία, στους εγκληματίες. Βέβαια και έχουμε ευαισθησία για αυτά τα πρόσωπα. Υπάρχουν πολύ σημαντικά που θα πρέπει να αναλάβουμε δηλαδή. Θα πρέπει να ε, τους παράσχουμε την ε, ανάλογη φροντίδα. Στέγαση. Αυτά ε, προσπαθεί να βάλει στο εναλλακτικό του ψήφισμα η πολιτική μας ομάδα. Δεν συμφωνούμε την έκθεση γιατί νομίζουμε ότι η, η εισηγήτρια ξεπέρασε τα ωραία τη εντολή τη και έκανε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν προ την εντολή τη Επιτροπή Γυναικών για το άσυλο, για την μετανάστευση και την επανένωση των οικογενειών. Όλα αυτά ε, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα τη έκθεση. Ε, οι θηλάουσε μητέρε, ε, οι έγκυοι μητέρε, οι δικέ του ανάγκε, αυτά είναι τα θέματα. Είναι πρόβλημα αυτό πάγιο Αντί να βοηθήσουμε, το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να αποδεικνύουμε πώ ξεπερνάμε την εντολή μα και ε, πώ υπερβαίνουμε τα αρμοδιότητά μα. Να το εμπόδιο στην εξέβρεση λύση. Συνάδελφοι, ε, παρακαλώ ψηφίστε το δικό μα ψήφισμα. Επόμενη μιλήτρια για 1,5 λεπτό η κυρία Μαρία Νόχελ, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάνιμπολ. Είναι εξαιρετική η έκθεσή της και έχει βάλει σωστά θεμέλια. Πρόκειται για την κατάσταση των γυναικών προσφύγων. Οι πρόσφυγες άνδρες και γυναίκες έχουν πολλά ίδια προβλήματα. Έχουν αυτό το φόβο να τους χωρίσουν από την ομάδα τους, το κρύο, ε, τις κακοχίες, την πείνα, την ανησυχία για το μέλλον. Όλα αυτά τα ζουν με τον ίδιο τρόπο άνδρες και γυναίκες όταν ε, είναι σε φυγή. Ε, αλλά οι γυναίκες έχουν επιπλέον προβλήματα. Συχνά συνοδεύονται από παιδιά για να μην πω ότι είναι και έγκυες πολλές φορές. Και επίσης πολλές φορές έχουν ξεφύγει από καταστάσεις στη χώρα τους όπου τους απειλούσε η βία ή ήταν εκτεθειμένες σε βία. Και στην προσφυγιά εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται με βία και από άλλους πρόσφυγες και με βία από ε, ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρέπει να τις βοηθήσουν αλλά και από άνδρες ε, στις χώρες στις οποίες ε, καταφεύγουν και πληρώνουν. Πληρώνουν το αντίτυπο όχι μόνο με χρήμα τους διακινητές αλλά και με το ίδιο τους το σώμα και μάλιστα μια τέτοια μέρα 8 Μαρτίου είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Πληρώνουν το τίμημα και με λεφτά και με βιασμό για να τους δώσουν ένα σωσίβιο και το μικρό τους κοριτσάκι τα ίδια για να πάρει το επόμενο σωσίβιο και λεφτά και βιασμό. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες πληρώνουν ένα πάρα πολύ ψηλό τίμημα όταν είναι πρόσφυγες και έχουμε ιδιαίτερα ευθύνη να προστατεύουμε τα γυναικόπαιδα ιδιαίτερα σε τέτοιε καταστάσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζούλη Γκέρλινγκ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας. Ούτε προσδοκεί στο να ζητήσει άσυλο. Καμιά γυναίκα δεν ξεκινάει ένα ταξίδι που θα καταλήξει σε ένα τόσο εκτρό αποτέλεσμα. Να σε χωρίσουν από το παιδί σου για λόγους βίας ή ασθένειας. Είναι τεράστια τα δεινά και ε, ο πόνος των γυναικών ε, προσφύγων. Έχουμε το καθήκον να τους προστατεύουμε από τη βία και το βιασμό και να τους δίνουμε υπηρεσίες υγείας και υποστήριξη. Αλλά η έκθεση νομίζω το παρατραβάει σε κάποιους τομείς. Ιδιαίτερα ε, ό,τι αφορά τη νομική αρρωγή και την οικονομική ε, συνδρομή. Άρα η δική μου αντιπροσωπεία Βρετανή συντηρητική θα υποστηρίξουμε το ΕΛΚ στο ψήφισμά του γιατί αναγνωρίζει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Εμείς κατανοούμε ε, τα όσα λέει η κυρία Χάνιμπολ και το πολιτικό ε, σκεπτικό και δεν θα καταψηφίσουμε την έκθεσή της. Η κυρία Βίξτρομ για ένα λεπτό παρακαλώ i brand och människor som inte haft samma tur som vi att leva i demokratiska välmående länder flyr för sina liv. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω πως στις χώρες που είναι δημοκρατικές και πλούσιες φτάνουν οι γυναίκες που εγκαταλείπτουν τις χώρες τους λόγω βίας και πολέμου. Ευχαριστώ την κυρία Χάνιμπολ για μια εξαιρετική έκθεση και όταν μιλάμε για θέματα τόσο σημαντικά όπως η κατανομή προσφύγων στις ευρωπαϊκές χώρες πολύ συχνά ξεχνάμε πως είναι ανθρώπινα όντα αυτά που κρύβονται πίσω από τους αριθμούς. Η έκθεση αυτή είναι εξαιρετικά ε, ισόρροπη και μιλά για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες. Δυστυχώς σήμερα ανησυχώ. Ανησυχώ για τα όσα προσπαθούν να προωθήσουν οι συντηρητικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτό ενδεχομένως θα χειροτερεύσει την τύχη αυτών των γυναικών προσφύγων. Δεν μπορώ να πιστέψω πως σήμερα, τη μέρα της γυναίκας, δεν θα δεχτούμε να καταδικάσουμε ε, αυτή την πίεση προς τις γυναίκες ε, πρόσφυγες. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να τους ε, στερήσουμε την αναπαραγωγική υγεία για να τις βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τα σεξουαλικά, τη σεξουαλική βία που αντιμετώπισαν. Ο κύριος Σέκη, ένα λεπτό, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα κάνουμε μια υποκριτική συζήτηση. Αν δεν παραμείνει ανοιχτή η Βαλκανική οδός είναι υποκριτική λέγω η συζήτηση αν δεν ακολουθήσουμε τις συστάσεις αυτές αλλά να ακούσουμε τα ακροδεξιά κόμματα. Ότι λέει να προστατεύουμε τα σύνορα και με ένοπλη βία και τα αφήνουμε να ακούγονται αυτά και δεν αντιδρούμε. Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών είναι απαράδεκτη. Βία με ένοπλη απέναντι σε γυναικόπαιδα έτσι θα θάψουμε την ευρωπαϊκή ιδέα. Η Ευρώπη θα πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη με τις γυναίκες και τα παιδιά πρόσφυγες και να αφήσουν με ανοιχτά τα σύνορα για αυτές τις ομάδες και να πούμε στους δεξιούς λαϊκιστές και ε, δεξιούς εδώ μέσα ότι θα μας βρουν απέναντι. Αυτό το οφείλουμε και στην Ευρώπη και στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Αυτά πρέπει οπωσδήποτε να το πούμε για να προχωρήσει η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Χάιντι Χάουταλα, για ένα λεπτό. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Χάουταλα. Απαντώντας, να συμφωνήσω με όσους ευχάριστησαν την κυρία Χάνιμπολ για την πλήρη της έκθεση. Βεβαίω, να λάβουμε υπόψη ότι κάποιοι θεωρούν ότι την εντολή τη, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα τα δικαιώματα τη γυναίκα. Αν ρίξουμε μια ματιά στην κατάσταση που διέπει αυτές τις γυναίκες στις απειλέ, στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, ε, θα πρέπει τότε να μπορέσουμε να του δώσουμε κάποιε εγγύσει για τα όσα χρειάζονται. η αναπαραγωγική υγεία θα πρέπει να προσεχτεί. Να το λάβουμε αυτό υπόψη. Θα πρέπει οι ευάλωτες ομάδε να προστατευτούν. Γιατί πρόκειται τώρα για μια τέτοια σημαντική ευάλωτη ομάδα. Η κυρία Νίβλερ για μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Καλό είναι που σήμερα την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας συζητούμε για την κατάσταση των προσφύγων γυναικών. Αλλά καλό θα ήταν, μάλλον και καλό ήταν που συζητήσαμε την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη προηγουμένως. Διότι πολλά από ε, τα όσα ισχύουν για τις γυναίκες πρόσφυγες και σωστά ζητούμε ως προστασία ισχύουν για όλες τις γυναίκες και θα πρέπει να τα ζητούμε και να τα εξασφαλίζουμε. Πρώτον, η βία κατά των γυναικών είναι απόλυτο ταμπού η σεξουαλική παρενόχληση, οι επιθέσεις, η βία, ο βιασμός θα πρέπει να τιμωρούνται αμήλικτα σε ποινικό επίπεδο και με περιφρόνηση να αντιμετωπίζονται με προστασία ε, ε, των θυμάτων ε, να προχωρούμε και όχι προστασία των δραστών. Επίσης θα πρέπει να σπάσουν τα κυκλώματα που διακινούν ανθρώπους. Αυτό χρειάζεται να μας βρει απέναντι και Βεβαίω αυτό αφορά γυναίκες πρόσφυγες, αλλά αφορά και πάρα πολλέ άλλες γυναίκες που δεν είναι πρόσφυγες. Έχουμε επανειλημμένα ασχοληθεί με το θέμα τη αναγκαστική πορνείας εδώ και τη διακίνηση ε, γυναικών για τέτοιου σκοπού. Ελπίζω να έχουμε αποτελέσματα στην Οδοκορυφή με την Τουρκία για να καταπολεμήσουμε τη λαθρομετανάστευση και να δημιουργήσουμε ασφαλείς νόμιμες οδούς με καταχώρηση και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για να έχουμε και πάλι τακτοποιημένες διαδικασίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα υποστηρίξω το εναλλακτικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Φυσικά. Ο κύριος Παντζέρη, παρακαλώ, για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρα από τα ιδεολογήματα και τις ανοησίες του εθνικισμού. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανταπόκρισή μας σε αυτή την πρόκληση θα είναι η απόδειξη κατά πόσον είναι ζωντανό το ευρωπαϊκό όνειρο και αυτές οι αξίες που ευάζησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Μεσόγειο και στο Αιγαίο φαίνονται όλα αυτά. Θα πρέπει να γίνει διαχείριση αυτής της κρίσης ε, δεν θα πρέπει αυτό να γίνει η αρχή της ακύρωσης της ε, ολοκλήρωσης. Χρειάζεται αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Επομένως, η μεταχείριση των γυναικών ε, και των ανηλίκων χρειάζεται να γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ ευάλωτοι σε αυτό το ταξίδι, γιατί τους εκμεταλλεύονται, υφίστανται σεξουαλική βία και κατόπιν ζουν μέσα στην τροπή και στο ψυχικό τραύμα που έχουν περάσει Άρα θα πρέπει να προσχωρήσουμε στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Οπότε θα πρέπει να ληφθούν και για το δίκαιο των προσφύγων ε, ε, η διαφορά των δύο φύλων και οπότε θα πρέπει να καλύψουμε, να κάνουμε αυτά που λέει η έκθεση Hannibal, να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε οξυδερκοί, στο βλέπουμε μακριά, να δείξουμε αυτή την αλληλεγγύη και κυρίως να έχουμε μια πολιτική για και ένταξη στην κοινωνία και στην οικονομία αυτών των ευάλωτων ε, προσφύγων. Θα πρέπει με πιο πολύ αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, κύριος Αρνέ Γκέρικε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε την κατάσταση των γενικών προσφύγων και του σώνα άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί συνάδελφοι συζητάνε σε ένα λεγόμενο πράσινο τραπέζι. Δηλαδή, τζογάρων. Κοιτάξτε κυρία Χάνιμπολ, πέρα από τη μύτη σας πριν ε, κάνετε τέτοιες εκθέσεις για το Κοινοβούλιο με λάθος εστίαση. Η Μεγάλη Βρετανία το τελευταίο έτος πήρε 166 σύρους πρόσφυγες. Δεν το επικρίνω, εντάξει, καλά κάνει. Αλλά μη φαντάζεστε τι γίνεται σε άλλες χώρες και μπορείτε να ε, πείτε σε άλλες χώρες τι να κάνουν με τις γυναίκες πρόσφυγες. Εμείς έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ε, ε, εθελοντές, 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες και η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν αναλάβει τεράστιες ευθύνες. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα και παγκόσμιο θα έλεγα. Συζήτησα χθε με εθελοντέ στην ε, δική σας έκθεση και η απάντηση είναι για πηγαίνετε σε ένα καταβλισμό μία μέρα να βοηθήσετε και δεν πρόκειται να ξαγράψετε τις ανοησίες. Και σας συνιστώ να ψηφίσετε αύριο όλοι το εναλλακτικό ψήφισμα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Επόμενος Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Χάνιμπολ για μια πολύ θαραλέα εισήγηση. Δυο φορές θύματα είναι οι γυναίκες πρόσφυγες και αντιμετωπίζουν κάθε είδους βία. Η ερώτηση είναι το εξή. Εκτός κοινοβουλίου θα μας ακούσει κανείς. Θα μας ακούσει το Συμβούλιο, θα μας ακούσουν τα κράτη-μέλη. Φοβάμαι πως μετά από την επέσχυντη συμφωνία με την Τουρκία δεν θα εισακουστούμε, γιατί κλείνουν τις πόρτες σε ανθρώπους που υποφέρουν και θέλουν μόνο να επιβιώσουν. Ίσως να γυρίσουμε πίσω και να θυμηθούμε τι έγινε το 39, όχι πριν από τόσα πολλά χρόνια. Η Ελίζα Μπεθέιτεμπεργκ στην Έλληνα, στο νότο της Γαλλίας, ε, έφτιαξε ένα βρεφοκομείο για να δεχθεί τις γυναίκες πρόσφυγες από την Ισπανία που εγκατέλειπαν την Ισπανία του Φράνκο που πέθαναν από το κρύο και από τις κακές συνθήκες και ε, στο ίδρυμα αυτό βρήκαν προστασία γυναίκες οι οποίες ε, εγκατέλειπαν τις χώρες τους γιατί αντιμετώπιζαν τις ναζιστικές θηροειδίες. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει. Ευχαριστώ. Η κυρία Αναμαρία Μαρία Κόρατσα Μπίλτ, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, όλο και περισσότεροι ε, ετούντες άσυλο είναι ετούσες άσυλο. Οι γυναίκες με παιδιά μόνε τους πολύ συχνά, οι γυναίκες και τα κορίτσια κινδυνεύουν να πέσουν στα χέρια διακινητών ε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και ακόμα και όταν είναι στην Ευρώπη. Η ασφάλεια και η ιδιωτική ζωή θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένε. Ξεχωριστέ υγειονομικέ εγκαταστάσει, πρόσβαση στην υγεία και την αναπαραγωγική θα πρέπει να είναι δεδομένη στι γυναίκε που το χρειάζονται. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κράτηση κοριτσιών ε, στις χώρους υποδοχής. Ε, θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους όταν γίνεται η συνέλευση για το άσυλο. Οι γυναίκες ε, έχουν υποστεί τραύματα, χρειάζονται υποστήριξη και ψυχολογική, όχι μόνο σωματική. Έχουμε κοινούς κανόνες. Ε, τα κράτη καλούνται τώρα να τα εφαρμόσουν με κατάρτιση για τους αστυνομικούς, για τις διοκτικές αρχές και άλλους για να καταλαβαίνουν ποια είναι τα θύματα ε, της βίας ε, με βάση το φύλλο και να τα προστατεύουν. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σχολείο. Για τα κορίτσια σχολείο σημαίνει δύναμη και συχνά και προστασία από την βία που η βία σε αυτή την περίπτωση είναι γάμος ανηλίκου με το στανιό. Ε, θα πρέπει οι πρόσφυγες και οι γυναίκες να εντάσσονται με τρόπο επιτυχή στη κοινωνία μας. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, Πρόεδρε, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να λέμε στις γυναίκες και τα κορίτσια που έρχονται στην Ευρώπη γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν από το πόλεμο ότι δεν είστε μόνες σας. Η Ευρώπη σημαίνει ασφάλεια για σας. Ας τις προστατεύσουμε και να βάλουμε την αξιοπρέπεια το, τέλος στο κέντρο της συζήτησής μας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει η Πρόεδρος, τώρα, λόγω του προκεχωρημένου της ώρας πρέπει να σας πω τα εξής δύο. Δεν θα δεχτώ μπλε κάρτες πια, σας είπα και προηγουμένως, και επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε τη δικασια Catch the Οι συνάδελφοι μίλησαν πάρα πολύ όλοι, εμακρηγόρησαν, δεν γίνεται. 12.30 έχουμε επίσημο προσκεκλημένο και 15 λεπτά για τις ψηφοφορίες, αλλιώς δεν θα προκάνουμε. Παρακαλώ να με συμπαθάτε. Η κυρία Κριστίν Βονταλόν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων της γυναίκας, θα πρέπει να πούμε στις γυναίκες πρόσφυγες που φεύγουν από τον πόλεμο και είναι τόσο ευάλωτες, ε, ότι ε, ξέρουμε ε, ότι είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε πλήρως στην πολιτική ασύλου το φύλλο. Χαιρετίζω το εξαιρετικό έργο της Μέρι Χάνεμπολ που στην έκθεση της λέει ποια είναι τα απαραίτητα εκείνα μέτρα για να προστατεύουμε τις γυναίκες και να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματά τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου. Γυναίκες και κορίτσια εφίστανται τα πάνδυνα ε, ε, αμήλικτο τρόπο και μαζί με τους ασυνόδευτους ανηλίκους κινδυνεύουν να πέσουν στα νύχια των διακινητών και των κυκλωμάτων. Αυτή η διαπίστωση μας θορυβεί και ζητεί περισσότερη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση ε, ε, της διακίνησης ε, των μεταναστών. Θα πρέπει επίσης να τερματίστη η κράτηση των ανηλίκων, των εγγύων γυναικών, των θυμάτων βίας και σεξουαλικής και των θυμάτων τράφικινγκ. Γιατί είναι που είναι οι άνθρωποι αυτοί τραυματισμένοι, θα επιδεινωθεί η κατάστασή τους με την κράτηση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γυναίκες πρόσφυγες και ΛΟΑΔ που μπορούν να υποστούν και χειρότερες διώξεις λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού. Είναι απαράδεκτη αυτή η βία που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια. Χρειάζεται ειδική προσοχή για την υποδοχή τους στην Ευρώπη με τρόπο ανθρώπινο και αξιοπρεπή. Είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτάχθηκε σε αυτό το κείμενο που είναι ε, παρόλα αυτά απαραίτητο για να καταδειχθεί αυτό που πολύ συχνά αποσιωπάται. Ε, κυρία Χέλγα Στέβενς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, παρά ε, τις καλές προθέσεις, η έκθεση Χάνιμπολ έχει χάσει το στόχο της. Συμφωνώ απολύτω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την κατάσταση τη δύσκολη που ζουν οι γυναίκες ε, και οι γυναίκες πρόσφυγες. Για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή που ζητάει ξεχωριστού κοιτώνε και ξεχωριστέ τουαλέτε ε, στα κέντρα υποδοχή για γυναίκε που είναι μόνε του ή μητέρε που ταξιδεύουν μόνε του με τα παιδιά του. Θα πρέπει κάθε μορφή βίας και βιασμού να ε, πατάσετε. Ε, βία κατά των γυναικών και παιδιών. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε και πρόληψη. Αλλά με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και των διάβλων ε, διέλευσης θα, χάσουν, θα χαθούν όλα τα προβλήματα αν ανοίξουμε τα σύνορα. Όλες οι γυναίκες πρόσφυγες χρειάζονται περισσότερη βοήθεια και περισσότερη νομική αρρωγή. Και πού είναι η αρχή της μη διάκρισης, απλώς και μόνο επειδή είσαι γυναίκα. Επίσης, στην έκθεση αυτή δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ ανθρώπων που ξεφεύγουν από τον πόλεμο ή από τα βασανιστήρια ή τις διώξεις και εκείνων που είναι οικονομικοί μετανάστες. Και κάτι άλλο. Οι ε, ανήλικοι που ζητούν άσυλο ε, δεν πρόκειται, λέει, να κρατούνται σε καμία περίπτωση. Άρα πρέπει να καταργηθεί αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία Υπάρχουν κάποιοι παράγρα, κάποιες παράγραφοι. Η πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο χρόνος σας έχει τελειώσει. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λευτέρης Χριστοφόρου. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, γιορτάζουμε σήμερα και απευθύνουμε όλοι ευχέ για την Παγκόσμια Μέρα τη Γυναίκα. Αλλά το ισχυρό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε ω Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι όσα λέμε σήμερα σε αυτή την επαιτειακή μέρα οφείλουμε ως ευρωκοινοβούλιο να τα εφαρμόσουμε και να τα καταστήσουμε πράξη. θεωρώ αξιέπαινη την πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αυτήν τη μέρα να τιμήσει όλος ιδιαιτέρως την πρόσφυγα γυναίκα γιατί στο μυαλό όλων μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή όλες εκείνες οι πρόσφυγες γυναίκες οι οποίες τριμώχνονται στους φράκτες της ντροπής για να μπορέσουν να σώσουν τις ζωές αυτών και τα παιδιά και των οικογενειών τους όλων εκείνων των προσφύγων γυναικών οι οποίοι ξεκινάνε το μακρύ ταξίδι της ζωής και του θανάτου για να γλιτώσουν από την καταστροφή του πολέμου όλων εκείνων των γυναικών πραγματικά που δίνουν τη μάχη των μαχών για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην προσφυγιά. όμως ταυτόχρονα δίπλα σε αυτές τις γυναίκες πρέπει να τιμήσουμε και την ελληνίδα γυναίκα που μπροστά στους φράχτες της ντροπής υψώνει τείχος ανθρωπιάς αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας στηρίζοντας και βοηθώντα τη γυναίκα πρόσφυγα στην ελλάδα στην ιδωμένη στα νησιά από άκρου άκρου όμως οφείλουμε σήμερα να τιμήσουμε και να αποκλειστούμε και στη γυναίκα της κύπρου. η γυναίκα της κύπρου είναι η πρόσφυγας γυναίκα της κύπρου η μοναδική ευρωπαία πρόσφυγας γυναίκα η οποία εδώ και 42 χρόνια δίνει τη μάχη για να επιστρέψει στις αιστείες της δίνει τη μάχη για να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που της τα παραβίασε η εισβολή και η κατοχή δίνει τη μάχη και την ελπίδα για να μπορέσει να ξαναζήσει ω άνθρωπο. οφείλει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να τιμήσει τη μοναδική ευρωπαία πρόσφυγα γυναίκα τη γυναίκα της κύπρου και την αγνοούμενη μάνα που περιμένει εδώ και 42 χρόνια για να βρει το παιδί της. Η κυρία Τόματσι τώρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. 38% είναι οι γυναίκες που το 2015 ζήτησαν άσυλο το εντάξει των όσων ζήτησαν ασυλό γιατί έτσι βλέπουμε ότι αυτά τα στοιχεία ε, επίσης λένε ότι έχουν γίνει αποδεικτές περισσότερες αιτήσει ασύλου ανδρών. Και βέβαια θα πρέπει κάτι να γίνει για τον πόλεμο αυτό στην Συρία, κάτι θα πρέπει να, γίνει με ντόπιε δυνάμεις Νομίζω ότι δεν κοινότητα πάντως. Αυτά τα στοιχεία δεν τα λαμβάνει υπόψη. Συνεχίζεται η χαλαρή πολιτική ασύλου και η πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Δεν θα πρέπει να μεταλλεύεται κανείς τη δυστυχία αυτών των ε, ανθρώπων και να προωθείται η άμβλωση. Όχι, δεν θέλω να κλείσουν τα σύνορα, δεν θέλω ούτε τα σύνορα να είναι μπάτε σκύλια λεύτερα. Σένφελτ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα γυναικόπαιδα που ε, φεύγουν ε, από τον πόλεμο και τη βία ε, είναι τραυματισμένα. Αλλά εδώ βλέπουμε το εξής παράδοξο. Πολύ συχνά ακριβώς αυτό που προσπαθούν να ξεφύγουν το βρίσκουν μπροστά τους καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και μάλιστα και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν φτάνουν εδώ. Καταλαβαίνω λοιπόν τα αιτήματα ε, της έκθεσης μεν, πλην όμως δεν συμφωνώ ναι. απολύτως με όλα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε αυτό το παράδοξο, να καταλάβουμε τους λόγους που παρατηρείτε, διότι πάρα πολύ συχνά στα κράτη-μέλη υπάρχουν θρησκείες, παραδόσεις, αρχές και αξίες που... Ε, ε, θεωρούνται υπεράνω του νόμου, του ευρωπαϊκού νόμου ή του εθνικού νόμου ή παράλληλα, εν πάση περιπτώσει, ή ε, γίνονται ανεκτά όλα αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι αυτοί που φτάνουν σε μια χώρα θα πρέπει να προσαρμόζονται και να συμμορφούνται προς την νομοθεσία και όχι το αντίστροφο. Αυτή είναι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου και η κοινωνία των πολιτών και θα πρέπει να ισχύει προς όλους εκείνους που έρχονται και καταφθάνουν στην Ήπειρό μας γιατί είναι προσκεκλημένοι μας. Θα πρέπει να υπογραφεί και η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης για το, το Συμβουλίο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σέντισχόφσκι και ζητώ συγγνώμη για την προφορά για 1,5 λεπτό. Eh, eh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, για την εξαιρετική προφορά σας στο όνομά μου. Αγαπητή Επίτροπε, όταν λέμε πρόσφυγας, οι περισσότεροι από εμά φανταζόμαστε έναν άνθρωπο 20 με 30 ετών που φτάνει στην Ευρώπη κινδυνεύοντας τη ζωή του για να επιτύχει το όνειρό του να ζήσει στην ευμάρεια την οποία μπορεί να παρέχει η ευρωπαϊκή κοινωνία σε αυτούς τους ανθρώπους. Λίγοι συνειδητοποιούν ότι σε αυτή τη φάση στην στα ελληνομακεδονικά σύνορα υπάρχουν τουλάχιστον, ε, μάλλον η μισή από τους πρόσφυγες είναι γυναίκες και παιδιά. Και αυτοί υπόκειται σε διακρίσεις. Στην ε, στην, στην αντιμετώπιση τους από τις αρχές. Διαρκώς τους επιτίθενται άντρες και οι γυναίκες αυτές ξεκινούν σε αυτή την πορεία όλο ένα και πιο συχνά και σε αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Ωστόσο η έκθεση αυτή έχει ευγενείς ε, προθέσεις και είναι κρίμα που το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει έχει πέσει θύμα μιας πολιτικής ε, σύγκρουσης, ε, έχει πέσει θύμα ε, στην επιθυμία να τοποθετηθούν εντός της ένα σωρό πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την κατάσταση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να το καταδικάσουμε και γι' αυτό στηρίζω το ψήφισμα του ΕΛΚ που παρέχει εναλλακτική. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Όπως ήδη είπα, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για τη διαδικασία Catch the Eye, διότι έχουμε τον προσκεκλημένο μας από το Ενίπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επειδή δεν έχουμε χρόνο και όλα τα σημαντικά και σοβαρά τα είπα στην ανεκτήρια ομιλία μου. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις σας, για τα σχόλιά σας και για την όλη συζήτηση και απλώς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα δραστικά μέτρα για να κάνουμε τη ζωή των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευκολότερη. Θα φροντίσουμε και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και όλες οι διαδικασίες ασύλου να γίνουν σεβαστές. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και για τη συντομία. Η συγκήτρια έχει το λόγο παρακαλώ η κυρία Χάνιμπολ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τα έχουμε πάει καλά ως τώρα και έχουμε σχετική ευημερία. Οι πρόσφυγες που αισθάνονται ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, τα σπίτια τους και τους αγαπημένους τους για να ξεφύγουν από την οδύνη και τον πόλεμο δεν βρίσκονται σε προνομιούχο θέση. Δεν βρίσκονται σίγουρα στη δική μας θέση. Ξέρετε πώς είναι κανείς ε, όταν εγκαταλείπει το σπίτι του, μόνο όταν είναι υποχρεωμένος το κάνει. Αυτή τη συζήτηση λοιπόν την κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι οι γυναίκες πρόσφυγες έχουν πολύ ειδικέ ανάγκες. Ανάγκες που τις εντόπισαν πολλοί από τους αγορητές. Θα σας παροτρύνω λοιπόν να καταψηφίσετε του ψήφισμα του ΕΛΚ, το οποίο αποδυναμώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που περιέχει το δικό μου ψήφισμα για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις ειδικές τους ανάγκες. Το ψήφισμα του ΕΛΚ αποδυναμώνει την επανένωση των οικογενειών, ένα ουσιαστικό ανθρώπινο δικαίωμα, την, ε, ε, τα δικαιώματα των εγγύων γυναικών, τη στήριξη για τις γυναίκες που έχουν υποστεί μορφές βίας και την ε, περίθαλψη των παιδιών μεταξύ άλλων, τη φροντίδα για τα παιδιά. Όπως υπόθηκε, τα δικαιώματα των γυναικών είναι δικαιώματα οικουμενικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια ιστορία και προστασίας των γυναικών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτή την οδό. Γι' αυτό σας παρακαλώ στηρίξτε τη δική μας ε, μορφή του ψηφίσματος. Ευχαριστούμε. Η συζήτηση ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή.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

Πριν, ε, αρχίσουμε, συνεχίσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τον ε, θάνατο της Έρτα Κάσερες που μας γεμίζει με οδύνη. Πρόκειται για μια αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία έχει, γεμίσει, έχει δώσει θάρρος ε, στην χώρα της γιατί αγωνιζόταν στην Ονδούρας για τα ε, δικαιώματα των ε, αυτοχθόνων. Η κυρία Κάσερες ήταν προσωπική γνώριμη πολλών από τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο. Για χρόνια είχε στενή συνεργασία μαζί τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει λοιπόν απερίφραστα το φόνο αυτό και καλεί την κυβέρνηση της Ονδούρας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει ο ή οι δράστες. Πιστεύω ότι το τραγικό αυτό γεγονός δεν θα αποθαρρύνει άλλους αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ότι θα τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους. Ιδιαίτερα στην Ανδούρας. Είναι πολύ εκείνοι οι οποίοι έχουν θυσιάσει τη ζωή τους στο βωμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Κάσερες, θα μείνει άσβηση στη μνήμη όλων όσοι τη γνώρισαν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Γκράντι, είπατε εκπρόσωποι και κυρίες και κύριοι, αρμοστή, συγγνώμη το ίδιο για τους πρόσφυγες κυρίες και κύριοι έχουμε σήμερα την ε, Διεθνή ημέρα της γυναίκας εορτάσει μέσα στο κοινοβούλιο φέτος όμως βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, κρίσης προσφυγικής και μεταναστευτικής που είναι μεγαλύτερη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και γι' αυτό αυτονόητο και λογικό είναι νομίζω αυτή την 8η Μαρτίου του 2016 να στρέψουμε ιδιαίτερα το βλέμμα και να αφιερώσουμε τις συζητήσεις μας στις γυναίκες τις οποίες πλήττουν αυτές οι κρίσεις. Από τον Ιανουάριο εφέτος έχει ξεπεράσει ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών που καταφτάνουν στην Ευρώπη εκείνων των ε, αρένων προσφύγων και ξέρουμε ότι οι γυναίκες σε αυτόν τον δρόμο εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους. Είναι πολλοί και πολλαπλοί οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται στο δρόμο της φυγής. Κάθε μέρα ακούμε τραγικές ειδήσει για τις διακρίσεις, για την προσβολή των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους, για την αφαίρεση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις γυναίκες. Είναι πολλές αυτές που βρισκόνται σε καταβλισμού προσφύγων και δεν ξέρουν εάν ή πότε θα μπορέσουν να βρουν και πάλι το δρόμο για μια αξιοπρεπή ζωή. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για μια αξιοπρεπή διαβίωση για κάθε γυναίκα στις πατρίδες τους, αλλά και αν χρειαστεί να φύγουν από αυτές τους στις χώρες προορισμού τους. Είναι πολλές οι θαραλέες γυναίκες που δεκαετίες τώρα αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών όπως η πρώτη πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας, η Σίμον Βέιλ. Για να αναφέρω ένα μόνο όνομα από τους δικούς μας, βουλευτές και πρόεδρος. Η παρακαταθήκη λοιπόν αυτών των γυναικών συνιστά ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Από την άλλη, τίποτε δεν είναι εγγυημένο επαόριστον. Και γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα να αγωνιζόμαστε για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Σε αυτή την έκθετη λοιπόν συνεδρίαση καλώς ορίζω τον Φίλιππο Γκράντι, είπα το αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Κύριε Γκράντι, είπατε αρμοστά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που με υποδέχεστε εδώ. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για τη Διεθνή ημέρα των γυναικών και τα δικαιώματά τους και να μιλήσουμε για το θέμα αυτό από την οπτική γωνία του οργανισμού, του οργανισμού για τους πρόσφυγες του παγκόσμιου του ΟΗΕ. Ε, Κυρίε και κύριοι, την περασμένη εβδομάδα ήμουν τη Λέσβο, το ελληνικό αυτό νησί, όπου ήταν την ελληνική ακτοφυλακή, να περισυλλέγει ε, ένα σκάφο με 200 ανθρώπους. Οι περισσότερες ήταν γυναίκες με παιδιά. Μερικά μικρή ηλικία, υπήρχαν κάποιε νεαρές γυναίκες, ηλικιωμένε και κάποιοι άρρωστοι άνθρωποι. Καθώς αποβιβάζονταν, τους μίλησα και άρχισαν να μου λένε ιστορίες. Ιστορίες από τις συγκρούσεις από τις οποίες δραπέτευσαν στη Συρία ή στο Αφγανιστάν. Τους κινδύνους του ταξιδιού τους και τις ανησυχίες τους για το τι μπορεί να τους επιφυλάσει το μέλλον ήταν ένα από τα πολλά παραδείγματα των σημερινών τάσεων μετακίνησης πληθυσμών παγκοσμίω. Πάνω από 60 εκατομμύρια ε, άνθρωποι παγκοσμίω έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την εστία τους. 42.500 άνθρωποι αναγκάζονται να αφήσουν τις εστίες τους καθημερινά. Η μισή από αυτούς τους ανθρώπους είναι γυναίκες. Παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εκτοπισμένων ανθρώπων, το 86% βρίσκονται σε άλλες επίρους, η Ευρώπη έχει πλέον αριθμούς ρεκόρ στις αφήξεις μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στις ακτές της. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το 2015 ένα εκατομμύριο άνθρωποι έφτασαν στην ε, Ευρώπη, διασχίζοντας τη Μεσόγειο, σε συνθήκες ε, ε, στις συνθήκες φουσκοθαλασσιάς ή με κάτι που δεν ήταν ασφαλή. Επίσης είδαμε τις εικόνες τους τις ελληνικές ακτές. Πάνω από 3.700 ε, ε, άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους. Αυτό είναι μια τραγική μαρτυρία για τη συλλογική μας αποτυχία να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Φέτος έως σήμερα 138.000 8.000 ε, μετανάστες και πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Νότια Ευρώπη. σύμφωνα με την κοινή γνώμη, η εικόνα που έχουμε είναι νεαροί ε, άνδρες ε, που φτάνουν στην Ευρώπη για να βρουν δουλειά. Όμως σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας θέλω να θυμίσω ότι αντιθέτως τα δύο τρίτα των ε, αφήξεων αυτών αφορούν γυναίκες και παιδιά. ήδη από την περσινή χρονιά στο 41%. Δείτε για παράδειγμα τη Φάτιμα, η οποία προσπάθησε να ξεφύγει από τον πόλεμο στη Συρία. Βρέθηκε σε κατάσταση σοκ στο λιμάνι της Σάμου είχε υποστεί τραυματική εμπειρία με βία που εξασκήθηκε εναντίον της από τους συνταξιδιώτες της. Πήγε σε νοσοκομείο για περίφαλψη και εκεί αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της της είχε εμπιστευθεί ε, αυτήν και την κόρη τη σε έναν άγνωστο για να ταξιδέψουν προ ένα ασφαλή προορισμό στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο άνθρωπο αυτό του έκλεψε όλα του τα ταξιδιωτικά έγγραφα, το κινητό και τα χρήματά του. Επίση, κακοποίησε τη Φάτιμα και δεν τη επέτρεψε να έρθει ξανά σε επαφή με το σύζυγό τη. Η Φάτιμα είναι μία από τι χιλιάδε γυναίκε και κορίτσια που κάνουν αυτό το ταξίδι μόνε του, προσπαθώντα να ξεφύγουν από τη βία και τι διώξει μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν παρόμοια μαρτύρια στην διαδρομή του προ την Ευρώπη. Έναν τόπο που περίμεναν και ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να βρουν καταφύγιο. Είναι πολύ απελπισμένοι παγκοσμίω που βλέπουν την Ευρώπη ω ένα τόπο ασφάλεια και ευημερία που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλωσορίζει του πρόσφυγε. Οι περισσότεροι δεν έχουν καλύτερες ή ασφαλέστερες εναλλακτικές και πολλές φορές προστρέχουν στους διακινητές τους, εμπόρους, με μεγάλου κινδύνου και ρίσκια. Να θυμήσω το σημαντικό γεγονό που συνήθω παραβλέπουμε ότι η ασφαλεστερες εναλλακτικε και πολλες φορες προστρεχουν στους διακινητε τους εμπορους με μεγαλους κινδυνους και ανθρώπων που συνηθω παραβλεπουμε οτι η πλειοψηφια των ανθρωπων που φτανουν στην Ευρώπη, το 88% προέρχονται από τις χώρες του κόσμου που βρίσκονται στο top 10 των χωρών που παράγουν μετανάστες. Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν, αλλά και Σομαλία επίσης. Αυτό είναι πραγματικά μια μετακίνηση προσφύγων, ε, κατά κύριο λόγο. Οι αριθμοί γυναικών και κοριτσιών μεταξύ του, διαρκώ αυξάνονται, όπω είπα, και πολλέ ταξιδεύουν χωρί του ε, άλλου ε, άντρε συγγενεί του. Βλέπουμε τον αριθμό εγγύων που φτάνουν εδώ, ή τι γυναίκε με μωρά και νεαρά κορίτσια και παιδιά που φτάνουν στην Ευρώπη. Μια πρόσφατη μελέτη του οργανισμού μα βρήκε ότι 20% των σύρων που φτάνουν στην Ελλάδα είναι οικογένειε που τις ε, έχουν αναλάβει γυναίκες χωρίς ε, συζύγους οι πατεράδε. Όπως η Φάτιμα, οι γυναίκες και τα παιδιά αυτά είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης πολλές φορές στα χέρια των ε, δίχως ενδιασμών εμπόρων οι οποίοι τις κάνουν να ταξιδέψουν από διαδρομές ανασφαλείς σε μέρη που δεν έχουν τις βασικές συνθήκες υγιεινής ή ασφάλειας όπως σε πάρκα, σε λεωφορεία ή σε συνδρομικούς σταθμούς ή στις, ε, στους αυτοκινητοδρόμους στην Ελλάδα βλέπουμε να αυξάνονται διαρκώς οι ρυθμοί προσφύγων και μεταναστών. Αυτή τη στιγμή περί πάνω από 35.000 βρίσκονται εκεί λόγω του κλεισίματος των συνόρων στα Δυτικά Αλβάνια δεν έχουν πλέον πρόσβαση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό έχει μια άμεση συνέπεια στις γυναίκες και στα κορίτσια, οι οποίες υποφέρουν δυσανάλογα και βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας. Εδώ λοιπόν με τους εταίρους μας πρέπει να στηρίξουμε τις τοπικές αρχές σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί και να βελτιώσουμε τις συνθήκες υποδοχής προσφέροντα ε, την βοήθεια και την αρρωγή που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να ε, αναχαιτήσουμε του κινδύνου και να βοηθήσουμε την ε, πορεία αυτών των γυναικών. Υπάρχουν πολλά σημεία και χώροι υποδοχή που έχουν ιδιαίτερε εγκαταστάσει για την υποδοχή των γυναικών και των παιδιών. Μαζί με τη UNICEF και την Διεθνή Κοινότητα του Ρυθμού Σταυρού έχουμε 20 ε, κέντρα για την υποδοχή οικογενειών και παιδιών, τα οποία είναι γνωστά και ω Blue Dots. Τα οποία προσφέρουν μέρημνα για γυναίκε και παιδιά που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε και πληροφορίε για τι επιλογέ του σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτά τα σημεία, αυτοί οι χώροι θα βοηθήσουν τι γυναίκε και τα παιδιά να μετακινούνται ασφαλέστερα ε, και να αντιμετωπίσουν τα τραύματα τη ε, κακοποίηση, τη εκμετάλλευση και τη εμπορία. Όμω, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, χρειαζόμαστε περισσότερα από ότι απλώ ανθρωπιστική απάντηση. Σε άλλε υπήρου, χώρε με λιγότερα μέσα από την Ευρώπη έχουν ανταποκριθεί σε πολύ μεγαλύτερε μετακινήσει πληθυσμών που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τι αιστείε του και συνεχίζουν να το κάνουν. Σε την ακριβών την αίθουσα παροτρήσεις ε, προς κράτη όλου του κόσμου να σεβαστούν τις αρχές για την προστασία των προσφύγων με τρόπο συντεταγμένο έχουν ακουστεί πολλές φορές και έχουν αντυχήσει τέτοιες όμως παροτρύνσεις ε, και εκκλήσεις αυτή τη στιγμή ισχύουν για την Ευρώπη. Αυτή η επίγουσα ανάγκη δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κρίση, πρέπει, μπορεί να τη διαχειριστούμε. Όπως γνωρίζετε χθε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνάντησε τους, ε, τον αρχηγό της Τουρκίας σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για να συζητούν το θέμα των προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Δεν συμμετείχαμε σε αυτές τις ζητήσεις και κατανοούμε ότι τις λεπτομέρειες ε, δεν τις έχουν αποσαφηνήσει ακόμα οι θύνοντες. Όμως μας απασχολεί πολύ σοβαρά οποιαδήποτε διευθέτηση θα περιλάμβανε την ε, τυφλή επιστροφή των διαφόρων μετακινούμενων από τη μια χώρα στην άλλη χωρίς να γίνονται σεβαστά τα ηχέγγια για την προστασία των προσφύγων και το διεθνές δίκαιο. Ένα ετών άσυλο θα πρέπει να επιστρέφεται σε μια τρίτη χώρα μόνον εάν την ευθύνη για την αποτίμηση της συγκεκριμένη αίτηση ασύλου επί της ουσίας την, μπορεί να την αναλάβει η τρίτη χώρα. Ο ετών άσυλο θα πρέπει να προστατεύεται από την ε, απομάκρυνση και θα πρέπει ως, σε ατομικό επίπεδο να μπορεί να λάβει όσα αναλογούν στους χρήζοντε προστασίας ασύλου βάσει των διεθνών προτύπων με πραγματική πρόσβαση στην εκπαίδευση, τη δουλειά, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική στήριξη που μπορεί να ε, χρειάζεται. Αυτές, αυτά τα ειχέγγυα θα πρέπει να καθιερωθούν νομικά με ένα μηχανισμό όπου η ευθύνη θα μπορεί να μεταφέρεται ε, με συγκεκριμένες συνθήκες για την αποτίμηση μιας αίτησης ασύλου. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει και μια ε, καλή εξέταση των αιτήσεων πρώτης αναχώρησης, ώστε να μην φτάνουν να γίνονται επιστροφές, ακόμη και αν πληρώνται οι άνωθοι προϋποθέσεις. Η Τουρκία ήδη υποδέχεται 3 εκατομμύρια πρόσφυγες, λίγο πολύ. Και είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα να μοιραστεί αυτήν την ευθύνη με τρόπο πιο σαφή. Καλωσορίζουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να προάγει την διαρκή υποδοχή προσφύγων σε σημαντικούς αριθμούς από όλες τις γειτονικές χώρες της περιοχής. Όχι μόνο από την Τουρκία και όχι μόνο Σύρους πρόσφυγες προς τις τρίτες χώρες. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί και ελπίζουμε ότι θα ισχύσει και για άλλες χώρες της γεωγραφικής αυτής ζώνης που έχουν στο έδαφος τους μεγάλο αριθμό προσφύγων όπως η Ορδανία και, και ο Λίβανος. Ε, πράγματι ε, ο Οργανισμός για τους Πρόσφυγες έχει καλέσει τα κράτη να ε, βελτιώσουν τους κανόνες τους για την υποδοχή ε, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουν σε ε, εμπόρους ε, ή δουλεμπόρους οι άνθρωποι σε επικίνδυνα ταξίδια. Θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες επανεγκατάστασης, της ανθρωπιστικής κατάστασης τους, της ε, προστασίας τους, της επανένωσης οικογενειών, καθώς και υποτροφίες για τους φοιτητές, αλλά και προγράμματα για την κινητικότητα των εργαζομένων. Θα πρέπει να προάγουμε τις δυνατότητες των σύρων ε, προσφύγων, όπως ε, προβλέπονται από τη Σύμβαση της Γενέβης. Εκεί θα συγκαλέσουμε μία σύνοδο υψηλού επίπεδου για να δούμε πώς μπορούν να κατανεμηθούν οι ευθύνε για την επανεισδοχή των σύρων προσφύγων. Εδώ τα κράτη θα κληθούν να αναλάβουν συγκεκριμένε χειροπιαστές δεσμεύσεις. Ελπίζουμε ότι το 10% των σύρων προσφύγων, του όλου αριθμού προσφύγων που αυτή τη στιγμή φτάνει τα 4,7 εκατομμύρια, θα μπορέσει να υποφεληθεί από αυτέ από αυτές τις διευθετήσεις. Επίσης, ελπίζω ότι οι πραγματικέ ροέ μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν με μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση. Βάσει τη αλληλεγγύη, βάσει τη πολιτική ηγεσία και βάσει τη κατανομή ευθυνών, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τι μετακινήσει των πληθυσμών και αποτελεσματικά την περασμένη Παρασκευή υποβάλαμε ένα σύνολο πρακτικών προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάτι μέλη τη, ώστε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Αυτές οι προτάσεις παραμένουν έγκυρες. Ε, επικεντρώνονται στο να βελτιώσουμε την καταγραφή και την εξέταση των αιτήσεων ε, των αφιχθέντων, ε, καθώς και τα προγράμματα επανακατάστασης στην Ευρώπη. Σημαίνει ότι η επανακατάσταση λειτουργεί και ότι τα απαραίτητα μέσα γίνονται διαθέσιμα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, προς την οποία εκφράζουμε την νομοσύνη μας. Πρέπει να εντείνουμε τις δυνατότητες απόκριση σε επίγουσες καταστάσεις στην Ελλάδα. Ο οργανισμός μας βρίσκεται εκεί με του υπευθύνους τους για να στηρίξουμε τι ελληνικέ αρχέ στην πράξη. Επίση, κοιτάζοντα το μέλλον, πρέπει να βασιστούμε στα μαθήματα που μόλι αντλήσαμε. Πρέπει η συμμόρφωση και η τήρηση των προτύπων του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου να γίνονται σεβαστά, ακόμα και σε στιγμές έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να ε, εμποδίσουμε την ε, απώλεια ζωών και την οδύνη των ανθρώπων αυτών, να προστατεύσουμε όσους κινδυνεύουν ιδίω τις γυναίκες και τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Αυτό συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες διάσωσης και έρευνας, την, τα συντονισμένα συστήματα για να προστατεύσουμε, να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τα ασυνόδευτα παιδιά και επίσης να έχουμε και μια αποτελεσματική απόκριση στην βία βάσει τη σεξουαλική ταυτότητα και του φύλου. Θα πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Όχι μόνο για να διαχειριστούμε αυτό την κρίση προσφύγων και μεταναστών, αλλά και για το μέλλον. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα συνεχίσουν να βαρύνονται με αυτό το δυσανάλογο άχθος για τις ανάγκες υποδοχής των προσφύγων. Η αλληλεγγύη που είναι τόσο καθοριστική σημασία σήμερα για την Ελλάδα και την Ιταλία ίσως να είναι κάτι προαπαιτούμενο και για άλλα κράτη στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι του Κοινοβουλίου, την επόμενη εβδομάδα σύγκρουση στη Συρία θα περάσει στον έκτο της χρόνο. Πάνω από 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι, όπως είπα, έχουν αναζητήσει άσυλο σε άλλες χώρες της περιοχής. 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ε, εκτοπιστεί εσωτερικώς μέσα στα σύνορα της Συρίας Υπολογίζεται ότι 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια άμεσα, μεταξύ των οποίων 4,5 εκατομμύρια σε περιοχέ που είναι δύσβατε. Με την πάυση των εχθροπραξιών για 10 ημέρε κιόλα, ε, ε, οι οργανισμοί του ΟΗΕ μαζί με τον δικό μα έχουν καταφέρει να παραδώσουν κάποια ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπου που έχουν υποφέρει από χρόνια πολέμου και στερήσεων. Εν τω μεταξύ στι γειτονικέ χώρε, παρά τη γενεοδορία των άλλων κυβερνήσεων και κοινοτήτων, οι Σύριοι πρόσφυγε αντιμετωπίζουν διαρκώ δύσκολε συνθήκε διαβίωση μετά από πέντε χρόνια στην εξορία. Μια πρόσφατη μελέτη που εκπονήσαμε με την Παγκόσμια Τράπεζα ανακάλυψε ότι στην Ορδανία και το Λίβανο 19% των Σύρων προσφύγων ε, ζουν κάτω από την εθνική γραμμή για τη φτώχεια, καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε νόμιμη εργασία και πολλοί δεν έχουν εξαντλήσει και όλα τους τα ε, περιουσιακά στοιχεία. Σε σύνοδο στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, η διεθνής κοινότητα δέσμευσε 10 δις ευρώ για δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες και που πρόκειται να βοηθήσουν και τις κοινότητες των χωρών υποδοχής για να βελτιώσουν τις δυνατότητες εκπαίδευση και διαβίωσής τους. Τα κράτη πρέπει τώρα να τιμήσουν αυτές τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη σύνοδο αυτή. Είναι κατεπίγουσα ανάγκη πλέον. Δεν μπορούμε να χάνουμε άλλο χρόνο για να σταθεροποιήσουμε τη συνθήκη διαβίωση των προσφύγων και των κοινοτήτων που του επιδόχονται στην περιοχή. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ελάχιστη ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί με την πάυση των εθνοπραξιών στη Συρία. Η Συρία όμω δεν είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που γνωρίζει κλειδονισμού. Από το 2015 η κλιμάκωση τη βία στο Ιράκ οδήγησε σε κύματα νέων εκτοπισμών. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια μόνο, περίπου 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλη τη χώρα. 16% ε, των ανθρώπων αυτών που φτάνουν στην Ευρώπη σήμερα είναι από το Ιράκ. Και σε τρει μόλι δεκαετία ε, οι Αφγανοί επίση παραμένουν ένα από του μεγαλύτερου ε, πληθυσμού προσφύγων ε, στον κόσμο. Με τουλάχιστον 6,2 εκατομμύρια καταγεγραμμένου πρόσφυγε. Οι περισσότεροι ζουν στο Πακιστάν και στο Ιράν. Όμω η αύξηση τη βία το δεύτερο μισό του 2015 προκάλεσε μεγάλου αριθμού εκτοπισμών πάλι μέσα στη χώρα και έξω από τα σύνορά τη και πολλά συνόδευτα παιδιά που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη ξεκίνησαν από το Αφγανιστάν. Σήμερα στο Αφγανιστάν ήταν 31 31 από 34 περιοχές πλήττονται από αυτοπραξίες με ένα εκατομμύριο ανθρώπους να έχουν καταγραφεί επισήμως ως εσωτερικώς εκτοπισμένοι και αύξηση κατά 78% σε σχέση με πέρσι. 25% των ανθρώπων που φτάνουν στην Ευρώπη είναι Αφγανοί και πολλοί χρειάζονται κατεπηγόντως βοήθεια. Αλλού στον κόσμο οι συγκρούσεις συνεχίζουν να ξεριζώνουν πληθυσμούς και να αναστατώνουν τις ζωές τους. Τα προγράμματα για τους πρόσφυγες στην Αφρική ακόμη δεν έχουν αρκετά κονδύλια. Ενώ ο αριθμός των πολεμικών συγκρούσεων και των εκτοπισμένων αυξάνονται διαρκώς. Νιγηρία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Νότιο Σουδάν και Μπουρούντι, για να αναφέρω μόνο μερικά παραδείγματα. Στο κέρας της Αφρικής έχουμε ένα θέατρο πολλαπλών εσωτερικών εκτοπισμών, ιδίως με Σομαλούς και σε πολλές από τις πιο έντονες περιπτώσεις εκτοπισμών στην Αφρική δεν μπορούμε να δώσουμε στους πρόσφυγες περισσότερα. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τους δώσουμε λιγότερα από τα ελάχιστα απαραίτητα για να επιβιώσουν. Κάποιες χώρες μάλιστα νομίμως δεν ε, τους επιτρέπουν να εργαστούν, οπότε η βοήθεια που λαμβάνουν είναι ελάχιστη στην Νοτιοανατολική Ασία, στην, ε, στον κόλπο της Μπεγκάλης, Πάνω από 3.000 μετανάστες και πρόσφυγες, κυρίως Ινδοί και Πακιστανοί, έχουν ανέβει σε σκάφη δουλεμπόρων ε, από πέρσι και πολλοί έχουν πνιγεί, μάλλον έχουν χάσει τη ζωή τους, όχι από πνιγμό όπως στην Μεσόγειο, αλλά από κακοποίηση στα χέρια αυτών των εμπόρων, από εγκατάλειψη και ασθένειες. Επίσης έχουμε ε, μια πολύ συγκεκριμένη κρίση προσφύγων στην Κεντρική Αμερική με χιλιάδες ανθρώπους από το Σαλβαδόρ, τις Ονδούρες και το Σαλβαδόρ που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις οργανωμένες και ένοπλες συμμορίες. Και πάλι όμως είναι Παγκόσμια Μέρα των Γυναικών και είναι ευκαιρία να θυμηθούμε ότι οι περισσότερες είναι γυναίκες και παιδιά έχουν χρησιμοποιήσει τις παραδοσιακέ παραδοσιακές οδούς μετανάστευσης για να αναζητήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο για το μέλλον τους. Όμως, ε, Κάποιοι είναι πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία, της διώξεις και τους εκβιασμούς. Σε ένα κόσμο λοιπόν όπου σοβούν ε, οι συγκρούσει, οι μαζικέ μετακινήσεις πληθυσμών είναι μια πραγματικότητα. Το να χτίζουμε τείχη και φράχτες για να τους εμποδίσουμε δεν είναι λύση. Απλώς θα αυξήσει την οδύνη των ανθρώπων αυτών που ήδη έχουν υποφέρει πολύ ε, σε βαθμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Οι γυναίκες παντού είναι οι πλέον εκτεθειμένες στον κίνδυνο. Ε, επειδή λοιπόν οι μαζικές μετακινήσεις και αφήξεις ε, δεν έχουν πάψει, πολύ συχνά η πρώτη αντίδραση των πολιτικών είναι να καταφύγουν στην, ε, ανά, στην στην χαραγώγηση, διότι το να προβάλλονται ψευδοεπιχειρήματα είναι τελείω ανεύθυνο. πραγματική απόκριση μπορεί να φαζείται στην αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κατανομή των ευθυνών και τον σεβασμό για το διεθνέ δίκαιο. Σήμερα γιορτάζουμε τα πολλαπλά επιτεύγματα προ το δρόμο για την επίτευξη τη ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική μα ζωή. Επειδή είναι η Παγκόσμια ε, ημέρα των γυναικών, να θυμίσω ότι την πρώτη φορά που γιορτάστηκε το 1975 ε, ή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να πετύχουμε την πλήρη ισότητα. Όμως και πάλι, να θυμίσω ότι είναι μια ευκαιρία σήμερα να θυμηθούμε ότι η διακριτική μεταχείριση και αποκλεισμή λόγω εθνότητας, θρησκείας και φύλου είναι μεταξύ των γενεσιουργών αιτίων που προκαλούν συγκρούσεις, διώξεις και ε, εξαναγκάζουν σε εκτοπισμούς. Σε 27 χώρες, για παράδειγμα, οι γυναίκες ακόμη δεν έχουν τα δικαιώματα με τους άντρες για να μπορέσουν να περάσουν την εθνικότητά τους στα παιδιά τους. Πολλές από τις γυναίκες που φτάνουν στην Ευρώπη έρχονται από αυτές ακριβώς τις χώρες, μεταξύ των οποίων Συρία και Ιράκ. Αυτό σημαίνει ότι οι πατεράδες δεν θα φτάσουν μαζί ή δεν υπάρχει, ή, ε, αν δεν υπάρξει πατρική, η συγκατάθεση του πατρός δεν θα έχουν εθνικότητα τα παιδιά αυτά, θα μείνουν απάτριδες, δεν θα έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και θα επηρεαστεί η δυνατότητά τους επιστροφής εάν το θελήσουν και το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως είπαμε και ακούσαμε, τα τελευταία 25 χρόνια το είπαμε επανειλημμένος. Δεν υπάρχουν πολιτικές λύσεις για τα ε, αίτια Ανθρωπιστικέ μάλλον λύσει για τα γενεσιουργά αίτια των ε, διώξεων και των συγκρούσεων. Ούτε για να αντιμετωπίσουμε στον πόλεμο τι μορφέ βία ε, και ε, τι διώξει σε πολλέ περιοχέ του κόσμου. Χρειαζόμαστε πολιτική δράση για να, για να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τα γενεσιουργά αίτια που προκάλεσαν τι συγκρούσει και να βεβαιωθούμε ότι άνθρωποι όπως η Φάτιμα και η μικρή της κόρη μπορούν να βρεθούν σε συνθήκε ασφάλεια χωρί να πρέπει να καταφύγουν σε εγκληματικά δίκτυα και οι οποίοι τι εκμεταλλεύονται. Αυτά δεν είναι αφηρημένα λόγια και έννοιες για τα οποία χρειάζεται να κάνουμε αφηρημένες δηλώσεις. Μιλάμε για πραγματικότητα, για γεγονότα ομά, τα οποία μόνο με τόλμη και πυγμή, με πολιτική ε, ανάληψη ευθύνη και, με, ε, αποφα... και με διορατικές πολιτικές αποφάσεις, καθώς και διεθνή συνεργασία, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και νέα έκφραση της ανθρωπιστικής μας θεώρησης, μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ε, η στιγμή η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των αξιών που διατείνεται ότι προσπίζεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Γκράντι. Εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο θα λάβει τώρα ο Επίτροπος Αβραμόπουλος. Αγαπητέ, είπατε ε, αρμοστή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα ε, και υπογραμμίσατε το θέμα των γυναικών μεταναστών και προσφύγων. Θα πρέπει να δούμε τους αριθμούς που φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα. Ε, συχνά, συχνά ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους. Οι ανθρώπινα όντα πολλοί από αυτούς είναι ευάλωτοι και χρειάζονται προστασία. Πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες τους παρά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Πολλές μητέρες κινδυνεύουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξεχνά και δεν ε, απεκδίεται των ανθρωπιστικών της ε, καθηκόντων. Πρέπει να ελέγξουμε τις ροές ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμες και να τις μειώσουμε. Ναι, χρειάζεται καλύτερα να διαχειριστούμε τα εξωτερικά μας σύνορα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κρατημέλη και τους πολίτες αυτών, αλλά και προσφέρουν των ανθρώπων που φτάνουν. Μάλιστα, χρειάζεται να σταματήσουμε τους διακινητές με τη βοήθεια της Europol που στέλνουν χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά σε έναν ε, πιθανό θάνατο. Ε, εκτός ε, είναι ευθύνη μας να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς για τους ανθρώπους που χρειάζονται νομική προστασία ώστε να μπορούν να έρθουν άμεσα νόμιμα και με ασφάλεια οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη και αυτό και συνεχίζω να καλώ τα κράτη-μέλη όχι μόνο να, να αποδώσουν όσον αφορά να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τον περσινό Ιούλιο για επανεγκατάσταση αλλά να δεσμευτούν και για περισσότερες ε, και γρήγορα Όλοι οι παράνομοι μετανάστες που φτάνουν από την Τουρκία θα επιστραφούν στην Τουρκία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό και νόμο, Διεθνή Νόμο. Για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ χρειάζεται να βελτιωθεί όμως η κατάσταση. Γι' αυτό και προτείνουμε ανθρωπιστικ... Ε, σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας για να χρησιμοποιηθεί εντός της Ένωσης και κατεπηγόντως χρειάζεται να προχωρήσουμε ε, σε μεγάλες κλίμακες ε, επανεγκαταστάσεις και να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τις δυνατότητες υποδοχής. Και για όλα αυτά ε, γνωρίζουμε ότι η υπατηρμοστία είναι ο σταθερός και απαραίτητος μας εταίρος. Προσβλέπουμε στενή συνεργασία με τον Φίλιππο Γκράντι, έναν άνθρωπο με προσωπικότητα που ήρθε στην ηγεσία της ΥΠΑ της Αρμοστία, σοβούσης της κρίσης, αλλά που είναι βετεράνος σε αυτά τα θέματα. Είναι άνθρωπος προσιλωμένος στο αιτήματα των προσφύγων και βασίζομαι στην πολιτική του βοήθεια. Καλωσορίζω λοιπόν και πάλι ε, την στενή συνεργασία που έχουμε θεσπίσει με την ΥΠΑΤΗΡΜΟΣΤΙΑ του ΟΗΕ και να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο της στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Η, η στήριξη της ΥΠΑΤΗΡΜΟΣΤΙΑ εκτιμάται ιδιαίτερα εντός και εκτός της Ευρώπης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πατερμοστία συνεργάζονται στενά για να βοηθήσουν την Ιταλία και κυρίως την Ελλάδα στην υποδοχή και την επανεγκατάσταση των μεταναστών. Ε, μαζί με την Πατερμοστία πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, ε, εφαρμογή του ανθρωπιστικού σχεδίου μαζί με την Τουρκία και να βοηθήσουμε για την υποδοχή των Συρίων στην Τουρκία. Όπως ξέρετε υπάρχουν δράσεις οι οποίες δεν περιορίζονται στα σύνορα της Ευρώπης. Το γεγονός ότι πάνω από 60 εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόσφυγες ή εσωτερικά εκτοπισμένοι σε ολόκληρη τον πλανήτη μας θυμίζει ότι θα πρέπει να ξεχνάμε πως η μετανάστευση δεν είναι μόνο θέμα της Ευρώπης, είναι παγκόσμια πρόκληση. Όλες στην, στη διεθνή κοινότητα θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους. Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να ανταποκριθούν στο αίτημα του ΟΗΕ για επαναγκατάσταση στις ε, περιοχές τους. Η διάσκεψη που οργανώνεται από την ΥΠΑ στις 13 Μαρτίου θα είναι η επόμενη ευκαιρία και χρειάζεται όλοι μαζί να σκεφτούμε πώς θα ανταποκριθούμε ε, θετικά σε αυτό το φαινόμενο που χαρακτηρίζει στην εποχή μας, στον κόσμο μας, στην κινητικότητα των ανθρώπων που αναμένεται να αυξηθεί μάλιστα για πολλούς και διάφορους λόγους και να πάρει διάφορες μορφές και να ακολουθήσει διάφορες δρόμους. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κινητικότητα του κόσμου. Ε, ούτε μπορούμε να τη σταματήσουμε. Χρειάζεται να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε χωρίς να αποσταθεροποιήσουμε τις κοινωνίες μας, αντιθέτως μετατρέποντας αυτές τις ροές σε μια αμφίδρομη ευκαιρία για τις χώρες υποδοχής και για τους μετανάστες. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι καθήκον της Ευρώπης και συμφέρον της να στηρίξει τους εταίρους που διαχειρίζονται τις ε, ροές και να ε, αντιμετωπίσει τις ρίζες αυτού του προβλήματος ε, των μετακινήσεων. Χρειάζονται λοιπόν σταθερές εταιρικέ σχέσεις, συνεργασία και με τρίτες χώρες αλλά και με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς. Σε μάλλα λόγια, χρειάζεται μια παγκόσμια στρατηγική σε αυτή την ε, πολυπρόσωπη και περίπλοκη κρίση των προσφύγων δεν μπορεί να υπάρξει μια ε, ομοιόμορφη προσέγγιση, ούτε να είναι ευθύνη μιας μόνο χώρας ε, ή ενός φορέα. Όλοι χρειαζόμαστε αλλήλους και χρειάζεται και να συνεργαστούμε. Γι' αυτό και η σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στην Ένωση και την τη αρμοστία του ΟΗΕ είναι τεράστια σημασία. Σε πολλή δουλειά μας περιμένουν τους επόμενους μήνες και ήδη είμαστε έτοιμοι και δεσμευμένοι να υλοποιήσουμε αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αβραμόπουλε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Γκονσάλες Πόνς τώρα. Είπατε, αρμοστή, η μέρα της ε, γυναίκας δεν είναι μόνο για τους, τα νούμερα, είναι για τα γεγονότα. Ε, σε πολλές χώρες του κόσμου, ωστόσο, οι γυναίκες έχουν λιγότερα δικαιώματα και λιγότερη ελευθερία. Αυτό είναι όντως ε, γεγονός. Οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ελευθερίες σύμφωνα με τον νόμο, αλλά όχι στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι γεγονός. Και εγώ ίδιος, αν ήμουν γυναίκα, θα ήμουν πολύ πιο... Θα είχα αντιμετωπίσει πολύ περισσότερε δυσκολίε στο να έρθω σήμερα εδώ να υπερασπιστώ την ισότητα των γυναικών. Ε, και αυτό είναι γεγονό. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι είναι αμφισβητήσιμη η χρησιμότητα εορτασμού τη ημέρα τη γυναίκα. Όμω είναι αναμφισβήτητο ότι υπάρχουν ένα σωρολόγιο χιλιάδε αίτια που ε- αιτιολογούν την ύπαρξη τη Διεθνού Μέρα ε, τη ημέρα. Υπάρχουν εκατομμύρια κορίτσια που δεν πάνε σχολείο επειδή είναι κορίτσια. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκε που δεν βρίσκουν δουλειά επειδή είναι γυναίκε. Και ένα ζωρό ηλικιωμένε που ποτέ δεν θα πάρουν σύνταξη γιατί είναι απλώ γιαγιάδε. Υπάρχουν γυναίκε που ε, κακοποιούνται, ταπεινώνονται ε, ακροτηριάζονται μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες και πολλές από αυτές είναι και φτωχές από πάνω. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3.500 γυναίκες ε, δολοφονούνται ε, κάθε χρόνο από άντρες. 8 κάθε μέρα, 8 σήμερα. Μία κάθε τρεις γυναίκες πάνω από, τις 60, από τα 60 έτη έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στη διάρκεια της ζωής της. Έχουμε λέμε και λέμε για τους Ταλιμπάν, αλλά και εμείς δεν είμαστε καλύτεροι εδώ πέρα. Ε, ε για κοιτάξτε τις ε, γυναίκες πρόσφυγες, τις πιο ευάλωτες που όχι μόνο υποφέρουν ε, από την ανισότητα αλλά και από τον πόλεμο που ξέρουν ότι Εκείνε πρέπει να αναλάβουν τα παιδιά όταν πρέπει να φύγουν και λόγω του συστήματος και της μαφίας ε, πέφτουν, πέφτουν και θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευση. Αυτές που έχουν λόγους για να φύγουν όπως ο ακροτηρισμό των γεννητικών οργάνων ή οι βιασμοί Ω ε, όπλο πολέμου στη Συρία το 25% των ανθρώπων που φύγαν ήταν ε, γυναίκε και παιδιά. Μπροστά σε αυτό το ανθρώπινο δράμα που ζούμε, οι λύσει που ακούμε, όλο ένα και πιο απάνθρωπε ακούγονται. Το να ορθώνονται τύχοι ώστε ε, τα γυναίκε με τα παιδιά να μην μπορούν να περάσουν, μα κάνει εμά, τους ίδιους να χάνουμε την ανθρωπιά μα, όχι εκείνε, Μια κοινότητα που δεν μπορεί να συγκινηθεί με μια γυναίκα που ζητά, ε, κάνει έκκληση για άσυλο με το παιδί της σε μια χαρτονένια κούνια, είναι μια απάνθρωπη κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν η δική μας κοινωνία. Το να είσαι γυναίκα, το να γεννηθεί κάποιο γυναίκα είναι μια κατάσταση. Το να στηρίξουμε τα δικαιώματα και τι ελευθερίε των γυναικών, ώστε να είναι ε, στην πράξη ίδια τα δικαιώματά τη στι ελευθερίε και στι ε, δικαιώματα των ε, ανδρών, είναι καθήκον μα, όχι μόνο για σήμερα, για όλη μα τη ζωή, αν θέλουμε να αξιοπρέπεια να αποκαλούμαστε Ευρωπαίοι. Σα ευχαριστώ κύριε Γκονσάρα Πόνς. Είσαι στο Δημοκρατική Ομάδα τώρα με την κυρία Γκίο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο καθένα καταλαβαίνει πλέον και ελπίζω τουλάχιστον ότι το αντιλαμβάνεται σε αυτήν την τωρινή κρίση. Οι γυναίκε πρόσφυγε, πολυάριθμε όλο και περισσότερο, αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Με την ευκαιρία τη Διεθνού ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών και με τη δική σας παρουσία κύριε είπατε Αρμοστά των Ηνωμένων Εθνών για πρόσφυγες θέλουμε ιδιαίτερα να μιλήσουμε για τις ανάγκες για διαφύλαξη της ζωής για επιβίωση των γυναικών αυτών θέλω να δώσω το λόγο στη Ρέμα σε μια νεαρή Σύρια και μεταφέρω τα λόγια της. Δεν μπόρεσα ποτέ να μπω στους καταβλισμούς να κοιμηθώ. Φοβόμουν ότι μπορεί κανείς ε, να με πλησιάσει και ε, να με θοπεύσει. Ήταν ε, ανάμεικτα τα καταλήματα, μεικτά τα καταλήματα. Δεν υπήρχε ασφάλεια. Έπρεπε να είμαι συνέχεια στον δρόμο για να μπορώ να κάνω ταξίδι. Πρόκειται για ένα, μια μαρτυρία λοιπόν, όχι μια γυναίκα που βρίσκεται στη Συρία, το Ιράκ ή οπουδήποτε αλλού θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την αυτονόητη μια ενδυμική βία. Εδώ στην Ευρώπη βρισκόταν η γυναίκα αυτή και ενώ μπορεί να φεύγει από ότι τη χώρα της για να αποφύγει τον πόλεμο πέφτει θύμα ή κινδυνεύει να πέσει θύμα των επιθέσεων. Αυτή λοιπόν ε, η ανησυχητική, η συγκλονιστική μαρτυρία της ΡΕΜ μας δείχνει ότι δεν έχουμε μπορέσει να δώσουμε απαντήσει Μπορεί η αναθεώρηση του πακέτου για το άσυλο να έχει βοηθήσει κάπω, αλλά παραμένουν ακόμη πολύ αδύναμες δυνατότητε μα. Ε, η Μαρία Ρεμό επίσης έχει πει ότι αυτέ οι επιθέσει κατά των γυναικών σημαίνουν ότι χρειάζεται προστασία σε κάθε στάδιο, με τη διαδικασία του ασύλου, με τι συνθήκες υποδοχής, με τα μέτρα ενσωμάτωσης, το προσωπικό ε, υποδοχή πρέπει να είναι καταρτισμένο, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής, ε, κοιτώνες, όχι μεικτοί ε, ως προς τα, τη σύνθεση των φύλων. Αυτά που μας λέει η ΡΕΜ με τη μαρτυρία της είναι ότι πρέπει πια να δράσουμε όλοι μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τους δεν μπορούν να επαναλαμβάνουν τη μία σύνοδο κορυφής μετά την άλλη χωρίς να λαμβάνουν μέτρα συγκεκριμένα για αποτελεσματική και συλλογική δράση για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής αλλά και ηθικής κρίσης την οποία έχει τώρα ε, βυθιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τα προβλήματα και πρέπει να δοθούν συγκεκριμένε απαντήσει. Πρέπει να βρούμε ασφαλέ καταφύγιο για να μπορούν να φτάνουν οι άνθρωποι χωρί να πέφτουν θύματα των διακινητών, οι οποίοι μόνο να πλουτίσουν σκέφτονται. Πρέπει να δώσουμε ε, λύσει με αλληλεγγύη ενδοευρωπαϊκή, μια ισότιμη, ε, έναν ισότιμο διαμοιρασμό των ευθυνών. Η Ιταλία και η Ελλάδα που έχουν κατακλειστεί και μόνο με το σταγονόμετρο 600 νομίζω την ημέρα μπορεί να φύγουν από τις χώρες αυτές. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις ως προς την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου που θα αλλάξει δραστικά αεκθεμελίων. Και επίσης πριν από μια πλήρη και συλλογική υλοποίηση του κοινού δικαίου του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί κανείς να δώσει απαντήσεις γιατί πια είναι σχεδόν ένα είδο λοταρία, λαχιοφόρου αγορά το ποιο θα μπορέσει να πάρει άσυλο στην Ευρώπη, όπω είναι η κατάσταση. Χρειάζεται μια ισορροπημένη, μια συλλογική λύση, η οποία θα ε, ενσωματώνει βεβαίω και το σεβασμό των υποχρεώσεών μα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επαύριο τη Συνόδου Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση με Τουρκία. Αυτή η διάσταση έχει ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία. Σα ευχαριστώ κύριε Αγγελιό, εκ μέρου ε, τη Ομάδα των Ευρωπαίων Στερετικών ο κύριο Κέρκοπ. Uh, uh, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είπατε εκπρόσωπε, κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για την ε, πρώτη προσφυγική κρίση με τη Βοσνιακή και είδαμε εκεί πόσα πράγματα, πόσα δεινά μπορεί να φέρει μια εμπόλεμη κατάσταση. Χαίρομαι που η δική μου η πατρίδα δεν έχει στρέψει την πλάτη ανώτη στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν όμως κάποιοι Ευρωπαίοι άνοιξαν τις πόρτες τους πέρσι σε, όσον, σε όποιους αναστούσαν μια καλύτερη ζωή, φαίνεται ότι έσπρωξαν προς τα πίσω μια σουρά που ήδη ήταν πολύ μακριά, εκείνους που είχαν πιο αδύρυτη ανάγκη για προστασία και υποδοχή. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι κίνδυνοι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ε, επιβίωσης, της διάσωσης στη θάλασσα, να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις που δεν θα ευνοούν τους διακινητές. Πρέπει να προσφέρουμε άσυλο, κοινωνική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή για να το κάνει αυτό πρέπει να αντιληφθεί ότι η επανεγκατάσταση και οι ελεγχόμενες προσφυγικές ροές είναι η μόνη λύση. Κύριε, ε, είπατε αρμοστά, ως ε, συντάκτης της εκθέσεως για την επανεγκατάσταση θα ήθελα να μπορώ να συνδυάσω το κείμενο αυτό με ένα φιλόδοξο ε, πρόγραμμα επαναγκατάσταση τη ΥΠΑ τη Αρμοστία μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τώρα το υφιστάμενο σύστημα δεν λειτουργεί. Α είμαστε ειλικρινεί, ορισμένα κράτη θεωρούν ότι του επιβάλλονται κάποιε λύσει και κάποια είναι διατεθειμένα να δεχθούν ορισμένο μόνο αριθμό. Δεν μπορεί να αποτελέσει αυτό λύση λοιπόν για μακροπρόθεσμη επιτυχία ενό συστήματο. Δεν θα δεν υποστηρίξουν κατά τρόπο αξιόλογο τα κράτη ένα σύστημα επανεγκατάσταση όσο δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί μεταναστευτικέ και προσφυγικέ ροέ. και βεβαίω όταν ο αριθμός των υποεπανεγκατάσταση. Όσο δεν υπάρχει λοιπόν σαφέ σχέδιο, όσο δεν υπάρχει ένα τέλο αυτή τη κρίση, μόνο να οξύνονται τα προβλήματα μπορούν. Μιλήσαμε για, προ... για δρόμους την Ευρώπη. Ευρώπη. Ναι, η επανεγκατάσταση μπορεί να το εξασφαλίζει αυτό. Μπορεί να προσφέρει ασφαλή μετάβαση για γυναίκε και παιδιά, στι οποίε με τόση, ε, τόσο εύκολο τρόπο αναφερθήκατε σήμερα. Να προσφέρει δηλαδή ασφάλεια σε σχέση με του απάνθρωπου αυτού διακινητέ. Είναι πολλέ οι γυναίκε που έχουν θύματα τη ε, εκμετάλλευση. Πολλοί είναι οι ανήλικοι, μη συνοδευόμενοι, για του οποίου έχουμε, τον οποίο έχουν χαθεί τα ίχνη αυτή τη στιγμή. Ε, θα μπορέσουμε λοιπόν να ελέγξουμε την κρίση αυτή και να προσφέρουμε ασφάλεια για τι γυναίκε και τα παιδιά αυτά με ένα σύστημα όμως το οποίο δεν θα πρέπει, θα πρέπει να είναι οργανωμένο. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να δείχνει και συμπόνια και να προσφέρει ασφάλεια, σταθερότητα στου πρόσφυγε και τι ευκαιρίε που πράγματι του αξίζουν. Σα ευχαριστώ, κύριε Κέρκοπ. Εκ μέρου των Φιλελευθέρων, η κυρία Βίξτρον. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Γκραντ για την τοποθέτηση και τις δηλώσεις σας. Αναλάβατε τα καθήκοντα, είπα του αρμοστή, κατά την χρονική εκείνη στιγμή κατά την οποία έφταναν ε, άνευ προηγουμένου προσφυγικέ ροές στις ακτές της Υπήρους μας. Δεν είχαμε δει τέτοια φαινόμενα τις τελευταίες δύο γενιές ε, και βλέπουμε και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις μεγάλες προκλήσεις ως προς τη στράτευσή μας, την προσήλωσή μας, την παροχή διεθνούς προστασίας για εκείνους που τη δικαιούνται. Τίνουμε στην Ευρώπη να λησμονούμε πως ζούμε όλο και περισσότερα χρόνια και ότι παραμένουμε με όλες τις δυσκολίες μας η πιο πλούσια ήπειρο στον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό η ίδια η καρδιά του συστήματος παροχής ασύλου αμφισβητείται από εκείνου που θα προτιμούσαν το δικαίωμα στο άσυλο να μην ήταν υποχρεωτικά χορηγούμενο δικαίωμα σε κάθε άτομο που το δικαιούται, αλλά μία χάρις η οποία θα απονέμεται κατά βούληση σε όποιον προτιμούσαν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και ο κίνδυνος λοιπόν να φτάσουμε στη στιγμή που κάποιος θα διαλέγει αν θέλει να, να προστατέψει, να προσφέρει προστασία σε πρόσφυγες και όπου κάποιοι θα έμεναν χωρίς προστασία με φρικτές συνέπειες. Μια φρικτή εικόνα όπου μια πλούσια δίκη, δύση θα αρνούνταν την παροχή προστασίας σε εκείνους που προέρχονται από χώρες αναπτυσσόμενες και θα τους έβαζε να καθόνται πίσω από τύχη ίσως στέλνοντας πότε πότε και μια επιταγή για να ισχυριστεί ότι τάχα φροντίζει τους πιο αδύναμους. Α, σε αυτήν την Ευρώπη εγώ δεν θέλω να συμμετάσχω. Και ως εκπρόσωπο της, ε, στα θέματα μετανάστασης εκ μέρους των φιλελευθέρων αλλά και μέλος της Επιτροπής για την αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου Κύριε Υπατέρμοστα, το μόνο μπορώ να σας μεταφέρω ως μίλημα για τους φιλελευθέρους και δημοκράτες ε, της Ευρώπης είναι ότι πάντοτε θα αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στο άσυλο. Όταν ορισμένοι εδώ στο σώμα ισχυρίζονται ακόμη ότι πρόκειται για μια επιλογή είτε μεν είτε δε. Δηλαδή είτε υποστηρίζουμε το θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα στο άσυλο, είτε υποστηρίζουμε τους πρόσφυγες. Όχι. Εμείς θα είμαστε το πλευρό σα και θα εξηγούμε ότι χρειάζονται και τα δύο αυτά στοιχεία για να λειτουργεί το σύστημα. Και παρεμπιπτόντω, η αρμοστία θα πρέπει να τύχει ακόμη περισσότερη υποστήριξη και όχι μόνο οικονομικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε σε εποχές γεμάτες προκλήσεις και δυσκολίες. Ας μην λησμονήσουμε όμως. Ας μην λησμονούμε ότι αυτή η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις ε, δυσκολίες αυτές. Σας βεβαιώνουμε λοιπόν ότι όλη η ομάδα μας θα είναι στο πλευρό σας σε αυτό το ε, άξιο έργο σας και, θα, ελπίζουμε ότι θα το φέρετε εις πέρας όπως και η άξιοι προκατοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα Ηνωμένα Έθνη, η ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, κρατάνε το κλειδί για την ε, πρόοδο του διεθνούς δικαιώματος στο άσυλο. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που ήρθατε σήμερα να μας μιλήσετε. Είναι όνειρο, πιστεύω, το ότι δεν κλείθετε να αναλάβετε περισσότερα καθήκοντα μέσα σε μια λύση ευρωπαϊκή για την αντιμετώπιση τη προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και οι προοπτικές υπάρχουν. Ναι, πρόκειται για μια παγκόσμια προσφυγική κρίση. Αλλά η προσφυγική κρίση δεν βρίσκεται εδώ στην Ευρώπη. Είπατε, μιλήσατε με τρόπο πολύ ευφύη, είπατε πολύ σημαντικά πράγματα. Σήμερα ιδιαίτερα μιλήσατε για τις γυναίκες που χρειάζονται υποστήριξη και προστασία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε αργότερα σήμερα να έγκρινε μια πολύ καλή έκθεση. Η Ευρώπη χρειάζεται να δεχθεί ακόμη περισσότερους και κατά τρόπο που θα σημαίνει ένα σωστό επιμερισμό των ευθυνών και των βαρών μεταξύ των κρατών. Δεν μπορούμε να κλείνουμε σύνορα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφαλή διέλευση. Να προστατεύουμε καλύτερα του ανηλίκου. Να βελτιώνουμε τα συστήματα κοινωνική ενσωμάτωση. Εχθέ επισκέφθηκε το καλέ τη Γαλλία και η κατάσταση την οποία διαπίστωσα εκεί δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελάτε παρακαλώ να δείτε το καλέ. Ελάτε να δείτε ποια κατάσταση έχει αναπτυχθεί εκεί. Είπατε ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η Ισλαμοφοβία και ο ρωτισμό στην Ευρώπη. Συμφωνώ απολύτω μαζί σας. Και εν δεν μπορεί να, αφήσουμε, να εγκαταλείψουμε την Ελλάδα στη μοίρα της, να αφήσουμε να μετατραπεί σε ένα τεράστιο καταβλισμό προσφύγων. Κύριε Γκράντι, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα διαπραγματεύεται με την ε, Τουρκία για να μην επιτρέπει στους πρόσφυγες να φτάνουν μέχρι εδώ, δεν αντιστοιχεί καθόλου με τις προτάσεις σας. Ξαναστέλνουν τους πρόσφυγες πίσω, μέσα στο ίδιο σκάφος με το οποίο φτάσαν στην Ευρώπη. Καμία σχέση αυτό με το προσφυγικό δίκαιο. Σα ευχαριστώ που το επισημάνατε. Με πολύ μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τιμά το προσφυγικό της δίκαιο και ελπίζω με τις δικές σας πιέσεις να δούμε κάποιες συγκεκριμένε αλλαγές προς το καλύτερο. Ο πρόεδρος εκ μέρους των Πρασίνων τώρα, τα ολόγω θα λάβει κυρία Χάρμς. Είπατε αρμοστά, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα χειροκροτήματα στο τέλος της ομιλίας σας, κύριε Γκράντι, απέδειξαν, νομίζω, ότι ιδιαίτερα τιμούμε το γεγονός ότι, φτάσατε, ότι ήρθατε σήμερα εδώ, ιδιαίτερο σήμερα εδώ, για να μα υπενθυμίσετε σε όλους μας εδώ στο σώμα τα προβλήματα, την κατάσταση αντίρρητης ανάγκης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα παιδιά σε αυτή τη μεγάλη και παγκόσμια προσφυγική κρίση. Ευχαριστούμε που μας συνταράξατε για άλλη μια φορά με, αυτό το, με, αυτό, την κλίση αφύπνισης ταυτόχρονα δείχνοντάς μας και με τα αριθμητικά στοιχεία ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Εμείς ως ευρωβουλευτές, κατά πλειονοψηφία τουλάχιστον, κατά πλειονότητα τουλάχιστον, αισθανόμαστε συγκλονισμένοι για το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει πια τόσο δύσκολο να τηρηθούν οι όροι της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες και την παροχή ασύλου. Βρισκόμαστε ενώπιον σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παρτίζεται από κράτη τα οποία έχουν όλα αναδυθεί ύστερα από πολέμους, καταστροφές, αποδιάρθρωση, αυτά που είχε δηλαδή ως ιστορία ο τελευταίος αιώνας και που θα έπρεπε να θυμούνται τι έχουν πράξει τα ίδια και τι έχουν υποστεί τα ίδια κράτη δεν μπορούν να αρθούν στο ύψος αυτής της παγκόσμιας κρίσης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η ομιλία σας είναι μια ομιλία που θα έπρεπε όλου να μας αφυπνίσει, όλου να μας ταράξει σε σχέση με τα όσα συζητήθηκαν εχθές με την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι βλέπουμε να γίνονται διαπραγματεύσεις με πολύ πολύ περιορισμένο οπτικό πεδίο. Ένα σύρος μπαίνει και ένα σύρος βγαίνει. Αυτή ήταν η απόφαση. Θα πρέπει αυτό να μας συνταράξει και συνδυαζόμενο με τα όσα ακούσαμε από εσά, κύριε Γκράντι γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η πρόθεση για εξασφάλιση της τάξης χάρη στην επανεγκατάσταση. Αλλά αυτή η μικρόψυχη προσέγγιση, ενώ ενός τόσο τεράστιου προβλήματος, μας συγκλονίζει. Έχετε καταστήσει με την ομιλία σας σαφές ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να δουν το σύνολο της καταστροφής, όλο το φάσμα των προβλημάτων και αυτό δεν το έχουν πράξει ακόμα προσπαθούν να προφυλαχθούν από μια καταστροφή αλλά ίσως με τον τρόπο αυτό και να συμβάλλουν στην ένταση, στην όξυνση των κρίσεων και των καταστροφών ή μη τι άλλο στην άμεση γειτονία μας και τον ευρύτερο κόσμο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Χάρμς, έχετε το δίκαιο. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να καθίσετε χωρίς φασαρία στις θέσεις σας. Κύριε Πάξας, ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίστε στις θέσεις σας. Δεν τιμά αυτό τη συζήτηση. Περισσότερο μοιάζουμε με γήπεδο ποδοσφαιρικό πριν από το σφύριγμα του διαιτητή. Παρακαλώ καθίστε. Δεν συνεχίζω τη συζήτηση μέχρι ότου καθίστε όλοι στι θέσεις σα Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα και πάνω απ' όλα δεν τιμά τη σοβαρότητα της συζήτηση που διαξάγεται εδώ αυτή την ώρα. natürlich nur ein Zufall, dass das überwiegend Männer sind, die hier. Τυχαίο προφανώ το ότι μόνο άντρε είναι όρθιοι ανάμεσα στα έδρανα και δεν έχουν λάβει τι θέσει του ακόμα. Παρακαλώ, κύριε Πάξα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Κύριε Πατέκ, πρόσωπε. Είναι μεγάλη μου χαρά που σα βλέπω εδώ. Ελπίζω η Ευρώπη εν τέλει να καταφέρει να προβλέψει όλα τα απαραίτητα μέτρα Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να βοηθήσουν τους πρόσφυγες αλλά όχι να ανοίξουν όλες τις πόλεις, όλες οι πόλεις τις πόρτες τους για τους μετανάστες. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να καταλήξουμε στι σωστέ πολιτικέ αποφάσει όταν μπλέκονται οι πολιτικοί. Εδώ δεν χρειάζεται να συζητάμε τα αυτονόητα. Οι άνθρωποι που είναι πρόσφυγε, που έχουν τραπετεύσει από τι αιστείε του γιατί έχουν υποστεί πολιτική δίωξη, χρήζουν προστασία. Υπάρχουν όμω άλλοι που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Εσεί είπατε, εκπρόσωπε. Δεν χρειάστηκε να δεχτείτε στο σπίτι σας ε, τους πάντες και ανθρώπους απρόσκλητου. Πώς το ζητάτε αυτό από τους ευρωπαίου πολίτες. Γιατί θέλετε να συμπεριφερθούν διαφορετικά. Ας πάψουμε λοιπόν να συζητάμε και ας αναλάβουμε κάποια στιγμή δράση. Να προστατεύσουμε την Ευρώπη κάποια στιγμή και από, την, ε, από τους μετανάστες. Να προστατεύουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. Όχι να αγοράζουμε την υποστήριξη της Τουρκίας με αντάλλαγμα δισεκατομμύρια. Θέλουμε να προστατεύσουμε πρώτα τους δικούς μας πολίτες και θέλουμε να ε, μετεγκατασταθούν σωστά οι πρόσφυγες ε, μεταξύ των κρατών. Όμως δεν είναι αυτό η βασική μας ευθύνη. Τα γενεσιουργά αίτια των πολεμικών συγκρούσεων πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια που προκαλούν αυτές τις μετακινήσεις. Ακούγεται κάπως περίεργο όταν ε, για τόσα χρόνια βλέπουμε φωτογραφίες με χωριά που καίγονται στη μια ή την άλλη χώρα και μόλις κάψουμε τα χωριά προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς που τρέχουν να ξεφύγουν. μεταξύ των ανθρώπων αυτών που έρχονται στην Ευρώπη κάποιοι δεν έχουν πληγεί ποτέ από πόλεμο ή σύγκρουση. Ευχαριστούμε κυρία Σαλβίνη. Για την Ευχαριστώ κύριο Σαλβίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ υποκρασία, υποκρισία στο όνομα των γυναικών ε, και τις Ευρωπαίες και τις ε, ε, μη Ευρωπαίες. Τι σκέφτεστε ότι θα γίνει με την Τουρκία στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργό τη έλεγε ότι γυναίκε και άντρε θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο και κάτι τέτοιο θα ήταν παραφύση. Ενώ ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση έλεγε πριν δύο χρόνια ότι οι γυναίκε δεν πρέπει να γελάνε και να προκαλούν δημοσίω. Αυτό λοιπόν το σώμα πιστεύει ότι θέλετε να είναι σωστό να φέρουμε στην Ευρώπη ανθρώπους τέτοιου είδους, τέτοιο κόσμο, ε, πραγματικά μου προκαλείται λύπηση. Λύπηση πραγματική. Ε, ανθρώπους που λένε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να γελάνε και να προκαλούν δημοσίω. Η Τουρκία δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Δεν θα είναι και δεν θα γίνει ποτέ μέρος της Ευρώπης των δικαιωμάτων των πολιτών, κατά τη δική μου άποψη. Τα 3% δισεκατομμύρια να τα δώσετε στου Ευρωπαίους ανέργους και όχι στο τουρκικό καθεστώς και την κυβέρνηση που το χρησιμοποιεί για να κλείνει τι εφημερίδε και να τι ξανανοίγει όταν το βολεύει. Όταν τι βολεύει. Και καθόλου για του πρόσφυγε και μετανάστε. Να τα δώσετε αλλού. Δείτε την Ιταλία. Οι αριθμοί, είπατε εκπρόσωπε, λένε ότι πέρσι σε 80.000 αιτήσει πολιτικού ασύλου που υποβλήθηκαν στην Ιταλία, το λέω για να τα ακούτε εσεί εδώ στο σώμα, μόνο το 5% έγινε ε, αποδεκτό ω πραγματικέ αιτήσει πολιτικού ασύλου. Μόνο 5% δέντρων των αιτήσεων απορρίφθηκαν. Δεδομένου ότι μιλάτε για γυναίκε στην Ιταλία τον Ιανουάριο του 2016, 7.000 αιτήσει πολιτικού ασύλου ε, ήταν μόνο 10% από γυναίκε. Ήταν όλοι γυναίκε άντρε και ενήλικη και σε πολύ καλή υγεία. Σύρι, κάτω των 30. Σύριες γυναίκες δεν βλέπουμε ποτέ. Εκτός εάν θέλετε να, να μην καταλάβετε ότι υπάρχει ανεξέλεγκτη ισλαμιστική εισβολή στη χώρα μας και σε όλη την Ήπειρο. Και μία ερώτηση εν τέλει. Πόσο σας κοστίζει κύριε είπατε εκπρόσωπε, πόσο κοστίζει στον ΟΗΕ ο οργανισμό σας, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητοι αυτοί οι υπάλληλοι, πόσα, ε, χιλιά, πόσα από αυτά τα δις των κονδυλίων φτάνουν πραγματικά στους πρόσφυγες και πό, τι κάνετε για τους ανθρώπους που μπορεί να κοιμούνται Και τι κάνετε για τα ακριβά ξενοδοχεία των υπαλλήλων ή τα ακριβά τους γραφεία. Τι κάνετε για τους Ευρωπαίους ανέργους, για τις γυναίκες που μπορεί να ανέργουν στην Ευρώπη, που μπορεί να πεινάνε και να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Το λόγο τώρα έχει ο μία εγγεγραμμένος βουλευτής, κύριος Φουντούλης. Κύριε Γκράντι, είστε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Δυστυχώς, όπως δείχνει η πραγματικότητα, μάλλον δεν τα πάτε και πάρα πολύ καλά στο έργο σας. Βεβαίως δεν είναι αποκλειστικά δική σας υπετιότητα, αλλά μάλλον και άλλων συναδέλφων σας στον ΟΗΕ. Εκείνοι οι συνάδελφοί σας που δεν αντέδρασαν στις και νεοαπικιακές πολιτικές των ισχυρών κρατών της δύσης που έχουν εισβάλει ή βομβαρδίσει σχεδόν το μισό πλανήτη. πού ήταν ο οηε όταν οι δυτικοί διέλυναν το αφγανιστάν τη συρία το ιράκ τη λιβύη την ουκρανία τη μισή σχεδόν αφρική και άλλες πολλές ακόμα χώρες; πού ήταν ο οηε όταν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όχι μόνο οι δυτικές φυσικά εκμεταλλεύονταν την εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να μπορούν να βγάζουν υπερκέρδη και να εξυπηρετούν το τέρας του υπερκαταναλωτισμού; όταν κράτη που τα θεωρούμε και προνομιακού μας συνομιλητές όπως είδαμε και στη χθεσινή σύνοδο γίνονται χορηγοί και υποστηρικτές των τούρκων που προστατεύουν την τρομοκρατία τους διακινητές και τους σύγχρονους δουλέμπορους. οφείλετε να δράσετε άμεσα οφείλετε να λάβετε μέτρα ώστε να σταματήσει η φωτιά του πολέμου που κατακαίει τη συρία και άλλες χώρες και οι μετανάστες να παραμείνουν στις πατρίδες τους για να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. οφείλουμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε τις ξεχωριστές ταυτότητες όλων μας τόσο τις δικές μας όσο και των χωρών προέλευσης για να μην δημιουργηθεί μια πολυπολιτισμική σούπα έρμεως στα χέρια των πολυεθνικών. όσον αφορά την πατρίδα μου η κατάσταση κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και περισσότερο απελπιστική πέραν από τις ευθύνες και τις ιδεοληψίες των κυβερνώντων που έχουν μπερδέψει τον ανθρωπισμό με την νομιμότητα και την ασυδοσία ποια είναι η αντίδραση του οηε τι έχετε κάνει ώστε να μην μετατραπεί η ήδη σκληρά δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση ελλάδα σε ένα απέραντο καταβλισμό. χορτάσαμε από λόγια και αναβολές δεν χρειαζόμαστε άλλα χρειαζόμαστε λύσεις και τις θέλουμε τώρα. δυστυχώς στην πράξη αποδεικνύεται ότι δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να μας προσφέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είπατε εκπρόσωπα, είπατε αρμοστά ε, για, τα θέματα των προσφύγων. Σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, ξέρετε, ο καθένας μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του. Οι δύο τελευταίες, δεν νομίζω ότι εκπροσωπούν επουδενή τα, τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Füge hinzu, ich füge και προσθέτω και προσθέτω Είπατε αρμοστά, προσθέτω κύριε αρμοστά, ότι σας ευχαριστεί θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο füge hinzu herr hoher kommissar ich ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και προσθέτω, είπατε αρμοστά, ότι σας ευχαριστούμε θερμά για την εξαίρετη ομιλία που εκφωνήσατε. Ευχαριστούμε εσάς και τους υπαλλήλους σας. Herr Coburn, Έχετε το λόγο κύριε Κόρμπαν παρακαλώ. Κύριε Κόρμπαν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω μόνο να ρωτήσω. εάν θεωρείτε ότι θα μπορούσατε ως πρόεδρος αυτού του καταπληκτικού σώματος να είσαστε ουδέτερος και να μην κάνετε παρατηρήσεις για αυτούς που βρίσκονται στην αποδόπλευρά του σώματος. Ε, Τελειώσατε. Τελειώσατε, ευχαριστώ, χαίρετε. Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό νομίζω ότι θα πρέπει να, παραμε... να διατηρείτε την ουδετερότητά σα. Θα ήταν αδιανόητη τέτοια συμπεριφορά στη Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν επιτρέπεται ο Πρόεδρος στη Βουλή των Κοινοτήτων να παίρνει το μέρος κάποιου. Κύριε Κόμπερν, ο υπάτος εκπρόσωπος, ο υπάτος αρμοστής των Εθνών ήρθε σήμερα σε μια εξαιρετική συνεδρίαση. Δεν είμαι διατεθειμένος να επιτρέψω να προσβάλλονται ο ίδιος και οι υπάλληλοι του και όταν εκδηλώνονται ρατσισμός, εγώ προφανώς θα αντιδρώ με μεγάλη ενεργητικότητα. Σας ευεβαιώ γι' αυτό.